Uh, λοιπόν, έπρεπε να ξεκινήσουμε στις 2.30, συνάδελφοι. Καθυστερήσαμε 10 λεπτά και ήδη έχουμε ξεπεράσει τα χρονικά όρια που είχαμε θέσει. Επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης για την απογευματινή συνεδρίαση. Η, η έκθεση πρωτοβουλίας για την κυβερνοασφάλεια και την άμυνα στον κυβερνοχώρο κύριο Πίτεν Τίμας, η σκιώδη συνεδρία στην προηγούμενη εβδομάδα και πολλέ συμβιβαστικέ ήδη έχουν αποτελέσει αντικείμενο συμφωνία. Είναι επίκαιρο το ότι ολοκληρώνεται τώρα αυτή η έκθεση. Στι τελευταία συνεδρία τη Επιτροπής μας πολλά σημεία συζητήσαμε, διάφορε πτυχέ ε, τη ε, Άμυνα στον κυβερνοχώρο. Τρει από αυτέ τι συζητήσει μπόρεσαν να επισέλθουν σε λεπτομέρειες και μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στις γενικές συζητήσεις για τη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα. Οπότε ενδείκνεται να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πέιτ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την όλη κατάσταση και πού βρισκόμαστε όσον αφορά αυτή την έκθεση. Έχετε το λόγο, ευχαριστώ. Όπως αναφέρθηκε, πράγματι έγινε με συνεδρίαση των σκιωδών. Αυτή η συνεδρίαση ήταν δημιουργικότατη, και διεξήχθη σε θετικότατη ατμόσφαιρα και το αποτέλεσμα το έχετε μπροστά σας και αύριο το πρωί στην ΑΦΕΤ θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. 30 συμβαστικές τροπολογίες έχουμε. Η έκθεση παρέχει την ανάγκη να δημιουργηθεί και να βελτιωθεί η αποτροπή στον κυβερνοχώρο και η προάσπιση ε, των ενόπλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να ε, προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Πολύ συχνά δέχονται κυβερνοεπιθέσει από άλλες χώρες και από μη κρατικού φορείς, ευρωπαϊκοί φορείς, οπότε θα πρέπει να αναπτύξουμε επιθετικές και αμυντικές δυνατότητες στον χώρο αυτό, ευρωπαϊκές. Όμως είναι όλο και δύσκολο να αντισταθούμε σε αυτές τις κυβερνοεπιθέσει σε επίπεδο κρατών μελών, λόγω τη φύση των επιθέσεων που δεν γνωρίζουν σύνορα και μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά το φαινόμενο και σε συνεργασία με του εταίρου μα και συμμάχου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει την πλατφόρμα για ευρωπαϊκή συνεργασία και να εξασφαλίσει έτσι ότι οι νέε προσπάθειε θα συντονίζονται στενά σε διεθνέ επίπεδο και εντό ε, τη ε, αρχιτεκτονική αμήνα τη διατλαντική συνεργασία με τον ΝΑΤΟ είναι ύψη τη σημασία και πρέπει να συνεχιστεί Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα, κρατών μελών, ανταλλαγή τεχνογνωσία, ανάπτυξη ευρωπαϊκών ασφαλών δικτύων για κρίσιμε υποδομέ και πληροφορίε. Θα πρέπει να βελτιωθεί επίση και η δύναμη τη ΕΝΗΣΑ. Μα λείπουν οι ειδικοί για τα θέματα ασφάλεια στον κυβερνό ασφαλεία ζητούμε να δημιουργηθεί έρασμος ε, στο θετικό τομέα και να γίνουν διάφορες προσπάθειες ανταλλαγή απόψεων. Χρειάζεται κατά τη εκπαίδευση, στην άμυνα, στον κυβερνοχώρο, να εκπαιδευτεί το θετικό προσωπικό όλων των ηλικιών, όλων των βαθμών και οι φοιτητέ όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό. Πρέπει να γίνουν κοινέ ασκήσει σε όλα τα επίπεδα και σε ύψιστο πολιτικό επίπεδο επίση. Τόσον αφορά τι διεθνεί προδιαγραφέ και κανόνε, παραδεχόμαστε ότι διεθνέ δίκαιο ισχύει και θα πρέπει να εφαρμόζεται και στον κυβερνοχώρο. Όλοι ζητούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί στι τωρινέ και μελλοντικέ συζητήσει για τι προδιαγραφέ στον κυβερνοχώρο και θα πρέπει μαζί με τον ΝΑΤΟ η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτήσει κριτήρια και ορισμού για τι κυβερνοεπιθέσει. Αύριο το πρωί, όπω σα είπα, θα ψηφιστεί έκθεση στην ΑΦΕΤ και ελπίζουμε ότι τον Ιούνιο στην Ολομέλεια ότι θα διεξαχθεί η τελική ψηφοφορία για μία ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, για τις συνεισφορές σας. Πάνω από 300 τροπολογίες λάβαμε. Για μία ακόμη φορά ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, τους κοιόδης εισηγητές, για την αποτελεσματικότατη αυτή συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα όπως έχουμε στην παράδοσή μας, α, είμαι σε θέση να δώσω το λόγο στον κύριο Λόπες Στόρες Βάιτ, τον εισηγητή του ΕΛΚ, αφού τον αφήσω να πάρει μια ανάσα και να βρει τη θέση του. Ευχαριστώ. Λόγω κυκλοφοριακού καθυστέρησα. Ξέρετε πώς είναι η κυκλοφορία στις Βρυξέλλες. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Πάες, τον ε, υπεύθυνο της έκθεσης, ε, που παρουσίασε και τις ε, τροπολογίες, που είναι πολύ καλή βάση εργασίας. Μας επέτρεψε να φτάσουμε σε καλές συμβαστικές τροπολογίες για να ψηφίσουμε αύριο. Θέλω να υπογραμμίσω κάποιες σημαντικές ιδέες κατά την απόψή μου ξανα, τις ξανακοιτάζω λιγάκι, τη συζήτηση που είχαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την στήριξη της ΕΝΗΣΑ θα πρέπει να ε, καθορίσει μια νέα αγορά για την κυβερνοασφάλεια και κυβερνοάμυνα. Θα πρέπει να τονίσουμε, τονώσουμε την συνεργασία για project ερευνητικά για να βρούμε κοινέ λύσεις για την κυβερνοασφάλεια και τους διάφορους τομείς, ε, ενέργεια, υγεία, μεταφορές, ε, οικονομικό τομέα και βεβαίως στην άμυνα. Ε, πολιτικές ε, τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο στρατιωτικό τομέα όπως, τομέα όπως τα drones, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά θα πρέπει να εγκριθούν Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να μείνει ουραγός, ε, αντίθετα, θα πρέπει να είναι προπομπό ε, σε αυτέ τι τεχνολογικέ εξελίξει. Εμεί ε, στο ΕΛΚ προτείνουμε να, χρησιμοποιήσουμε, να υπάρξει ένα, ε, μια πολιτική και στρατιωτική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει καλύτερο σχεδιασμό, οδηγίες οδηγίε και πραγματική και αποτελεσματική έλεγχη. Και μια αρχή για τον κυβερνοχώρο που θα είναι ένα σημείο που θα συνδέει τα κράτη-μέλη και Θα πρέπει να ε, συντονίσουμε την επιχειρησιακή δραστηριότητα των κρατών μελών, ούτω ώστε να φτάσουμε σε επιχειρησιακούς στόχους της κοινή πολιτικής ε, άμυνας και ασφάλειας στα πλαίσια της ε, ΠΕΣΚΟ. Μία κυβερνοαρχή, η οποία θα προωθεί την, την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών για να ανταλλάσσονται και πληροφορίες που είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Να συνδυάσουμε το πολιτικό και στρατιωτικό τομέα ε, για να καταλάβουμε καλύτερα τις απειλές στον κυβερνοχώρο και να αντιδρούμε καλύτερα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση ε, του νέου πεδίου μάχης που αντιμετωπίζουμε στο ίντερνετ. Θα πρέπει να δείξουμε και εντός και εκτός τις αμυντικές και επιθετικές μας ε, δυνατότητες. Τέλος, στα πλαίσια της κυβερνοάμυνας θα αντιμετωπίσουμε συνεχείς αλλαγές και είναι πολύ δύσκολο για τους νομοθέτες για μας να προλάβουμε τις εξελίξεις. Ε, συχνά κάποια συμβάντα δεν τα ξέρουμε, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τους μηχανισμούς για να προσαρμοζόμαστε και να τους επικαιροποιούμε. Τέλος, όπως είπα και στην αρχή, με τις συμφωνίες που πετύχαμε ε, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και συγχαίρω τον εισηγητή για όλη την προσπάθεια που έχει γίνει και για τις συζητήσεις που κάναμε. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Καθήκον μου να, να φορέσω το καπέλο μου της εισηγήτριας των σοσιαλιστών υπό αυτή την ιδιότητα θα μιλήσω, απηχώ και τα σχόλια του κ. Λόπες Εστορίας White. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Έξοχο το κείμενο, το αρχικό, το οποίο επεξεργαστήκαμε. Αυτό που επεξεργαστήκαμε σαν σκιώδη εισηγητέ, επεξεργαζόμενοι 300 τροπολογίες, που μας υπευλήθησαν. Όπως αναφέρθηκε, ευρία ήταν η υποστήριξη όλων των ομάδων όσον αφορά την προσέγγιση της Ευρώπης για την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Οι συμβαστικές τονίζουν ότι η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ είναι ουσιαστικό κομμάτι της άμυνάς μας στον κυβερνοχώρο της Ευρώπης. Ταυτόχρονα η άμυνα της Ευρώπης, η Ένωση Αμυντική της Ευρώπης χρειάζεται στρατηγική ε, αυτονομία. Ήταν και το άλλο θέμα. Ότι υπάρχουν κρατικοί και μη κρατικοί φορείς που αναμειγνύονται στις απειλές που απευθύνονται προς την ασφάλειά μας. Και είναι δύσκολο να βρει κανείς ποιος ακριβώς είναι ο επιτιθέμενος. Χρειάζεται επίσης και η ατοδικαστική ούτως υπήν προσέγγιση όσον αφορά αυτές τις επιθέσεις. Και χρειαζόμαστε κοινή θέση μετά από μια κυβερνοεπίθεση για να διαπιστώσουμε τα στοιχεία. Λοιπόν, και κάτι άλλο που είναι σημαντικό και υπογραμμίζει στην έκθεση η διεθνής κοινότητα πρέπει να συμφωνήσει όσον αφορά την εφαρμογή διεθνών προδιαγραφών στον κυβερνοχώρο. Και οι κακεντρεχείς επιθέσεις, οι κακόβουλες επιθέσεις είναι και παράνομες και δεν μπορούν να λαμβάνουν χώρα χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Η έκθεση αναφέρεται σε πολλά θέματα που συζητήσαμε στέντε πριν, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας, και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμπληρώνει το ΝΑΤΟ διατηρώντας στρατηγική αυτονομία. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η έκθεση θα συμβάλλει στη διεξαγωγή της συζητήσεως και θα δείξει ότι το κοινοβούλιο μας είναι σοβαρό. Θέλει να εξασφαλίσει το ότι η Ευρώπη είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την κυβερνασφάλεια και την άμυνα στον χώρο, τον κυβερνοχώρο. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο του. Και τώρα θα παρακαλούσα άλλους εισηγητές αν επιθυμούν, να λάβουν το λόγο. Δεν νομίζω ότι έχουμε εκπρόσωπο του ECR. Α, έχουμε. Ορίστε, υπέροχα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε με την αφετηρία αυτού του εγγράφου και με τις προθέσεις, γιατί η κυβερνοασφάλεια είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τη λειτουργία των υποδομών μας και της αμυνά μας συνολικά. Ε, έχουμε όμως κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με αυτά που είπατε, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την αυτόνομη λειτουργία της άμυνάς μας, ε, τα τρίτα των χωρών συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, τα τρίτα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται και πολιτικές προσπάθειες και υπάρχει και μια πολιτική προσθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η οποία θα πρέπει να βοηθήσει τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και να μην δημιουργήσει μια δεύτερη παράλληλη δομή, ένα δεύτερο παράλληλο πλαίσιο. Όταν υπάρχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες ε, αρμοδιότητες, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια επιδείνωση της άμυνάς μας και όσο σε μια βελτίωση. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα. Θέλουμε να συνεργαστούμε, ούτω ώστε όμως να αυξήσουμε την ασφάλειά μας και την κυβερνοασφάλεια. Έχουμε όμως κάποιες επιφυλάξεις ε, σε ό,τι αφορά αυτή την αυτονομία που θα οδηγούσε σε μικρότερη αλληλεγγύη ε, στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ απέναντί μας. Gracias, Presidenta θα παρουσιάσουμε μία μειοψηφική έκθεση. και δεν συμφωνούμε με την ουσία της έκθεσης. Έχουμε εντελώ διαφορετική αντίληψη. Δεν υποστηρίζουμε την ενιαία αγορά της κυβερνοασφάλειας, ούτε τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ για θέματα κυβερνητικής ασφάλειας. Και υπάρχουν και πολλές, πολλά κενά όσον αφορά ε, την ασφάλεια, την πολιτική ασφάλεια και τον περιορισμό των δικαιωμάτων των κρατών μελών και χρησιμοποιούνται κάποια μέσα ανεπαρκή θεωρούμε του πολιετούς πλαισίου. Γι' αυτό θα υποβάλουμε έκθεση μειοψηφική και θα καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η Ο Πράσινος Σκιώδης ε, συμμετείχε ιδιαίτερα στις των Σκιωδών, ο κύριος Τάραντ, αλλά δεν είναι παρόν τώρα. Ο κύριος Καστάλντο και ο κύριος Σαφχόζερ επίσης δεν είναι παρόντες. Οπότε κλείσαμε τη συζήτηση. Α, α εσείς παρακαλώ. Να κάνω μερικές σύντομες παρατηρήσεις. το σημείο αφετηρίας του εισηγητή. Ε, ε, διαρωτώ με αν ήταν σωστό. Υπευλήθησαν πάνω από 300 τροπολογίες. Αυτό δεν ε, αποδεικνύει ότι ήταν κακό το σημείο αφετηρίας, αλλά υπήρξε ανάγκη διεύρυνσης και συμπλήρωσης κάποιων θεμάτων, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα η κυβερνοασφάλεια. Είναι ένα θέμα που για πρώτη φορά στην πραγματικότητα σε βάθος συζητήθηκε για πρώτη φορά λοιπόν από εμά. Και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αύριο θα μας βοηθήσει. Θα έχουμε ένα καλό κείμενο. Το μόνο θέμα που με ανησυχεί είναι ότι καθυστερούμε. Έχουμε χάσει πολύ χρόνο. Και δεν θα προλάβουμε να καλύψουμε την καθυστέρησή μας σε θέματα ασφάλειας Γιατί γενικά Ιστερούμε, ολιγορούμε. Δεν αρκεί μόνο ε, η υιοθέτηση νομοθετημάτων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα τις απειλές που υφιστάμεθα. Αλλά πιστεύω ότι η έκθεση του συναδέλφου πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά Ορισμένε καταστάσει είναι ιδιαίτερα σοβαρέ και πρέπει να αντιδρούμε πολύ σύντομα. Αυτό λέγεται. Και τονίζουμε ότι η κυβερνοασφάλεια δεν είναι ε, θέμα μόνο κάποιων κρατών μελών. Είναι θέμα που μας αφορά όλους. Είναι θέμα της γενικότερης κοινή μας ασφάλειας. <clears throat> και να πω στον συνάδελφο ότι τον ευχαριστώ πολύ και είμαι πεπισμένο ότι θα είναι θαυμάσια η έκθεσή σας. Ευχαριστώ όλοι, πρόεδρος. Κύριε Πέτ, θέλετε να επανέλθετε. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Για τη συνεργασία Ένωσης ΝΑΤΟ για την κύβερνο άμυνα είναι φανερό ότι πρέπει να υπάρξει και επανειλημμένα έχει τονιστεί στο κείμενό μου. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ μέλη της Ένωσης και του Μπαλίν. Και τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, της κυβερνοάμυνας είναι πολύ σοβαρά. Αντιμετωπίζουμε πολλές απειλές. Άρα θα πρέπει να ενταχθεί η κυβερνοασφάλεια στη γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και των κρατών μελών. Έτσι δεν υπονομεύουμε την Ένωση ή τον ΝΑΤΟ ή τη συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές διαταράξεις, ελαφρές διαταράξεις στις σχέσεις Ένωσης ΝΑΤΟ. Ναι βεβαίως υποβλήθηκαν πάνω από 300 τροπολογίες. Αλλά επενθυμίζω ότι πριν ξεκινήσει η εκπόνηση της έκθεσης κάναμε μια συζήτηση όπου είπαμε ποια θα πρέπει να είναι τα όρια και η αρχιτεκτονική του κειμένου και είπαμε ότι πρέπει να επικεντρώσουμε στην κυβερνό άμυνα να μην θίξουμε όλες τις πλευρές της κυβερνοασφάλειας που είναι πολύ ευρύτερο θέμα εντάξει μπορεί να συμφωνεί να διαφωνεί κανείς αλλά έτσι αποφασίστηκε τότε και γι' αυτό πολλοί συνάδελφοι υπέβαλαν τροπολογίες που διευρύνουν κατά πολύ το πεδίο της έκθεσης σε σχέση με την αρχική μας αντίληψη. Και αυτό δημιουργεί κάποιες συγχύσεις. Γιατί ξέρετε, πολλοί δεν κάνουν ε, σαφή διαχωρισμό αυτών των δύο. Μαζί με τους κοιόδης. Λοιπόν, φυσικά επιχειρήσαμε και νομίζω και επιτύχαμε να επιτύχουμε αυτήν την ισορροπία μεταξύ την γραφειοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων ποιος θα πρέπει να πάρει δηλαδή τις αποφάσεις και μετά την ουσία του θέματος. Συγγνώμη βεβαίως που δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω όλες τις καλές ιδέες των συναδέλφων γιατί δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν με το πλαίσιο που είχαμε καθορίσει. Ευχαριστώ πολύ και να δούμε τι θα γίνει και στην ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για όλη σας τη δουλειά. Και τον καλό τρόπο αντιμετώπισης του επίκαιρου αυτού θέματος. Λοιπόν, όπως ήδη υπόθηκε, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στην ΑΦΕΤ και στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Οπότε, το επόμενο θέμα στη μέση διάταξη και την κατάλληλη στιγμή μάλιστα, διότι έχουμε τη δεύτερη εξέταση της έκθεσης του κυρίου Πάσκου για τις σχέσεις ε, Ένωσης ΝΑΤΟ ιδιαίτερα για να συζητήσουμε τις τροπολογίες και τις συμβαστικές. Ο κύριος Πάσκου εξεπώνησε μια αναλυτική εκθέση που καλύπτει όλες τις βασικές πλευρές της εξελισσόμενης αυτής σχέσης. Υποβλήθηκαν 360 τροπολογίες, έγιναν ε, αναλυτικές συζητήσεις. Οπότε να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Πάσκου. Θα φτάσουν ε, τα 45 λεπτά, κυρία Πρόεδρε, για να παρουσιάσω όλα τα σημεία. Όπως αναφέρατε, είχαμε 360 τροπολογίες και καταλήξαμε σε 22 συμβαστικές τροπολογίες, ευρέως υποστηριζόμενες από όλα τα μέλη. Προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε τη συνοχή και το πνεύμα της ε, έκθεσης. Όλοι γνωρίζουν ότι κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένος με την τελική εκδοχή της εκθέσεως. Ε, αλλιώς δεν θα είχαμε έκθεση. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που δεν συμπεριελήφθησαν, διότι κάποιες από τις ιδέες που περιείχαν είχαν ήδη αναφερθεί με κάποιο τρόπο στην έκθεση άλλες είναι πολύ λεπτομερείς, έτσι δεν υπάρχει περιθώριο να γίνουν αποδεκτές, δεν υπάρχει χώρος. Άλλες τροπολογίες είναι εκτός θέματος. Εν γέννη, η συνεργασία ήταν καλή μεταξύ των σκιωδών. Δεν διαβλέπω κάποια σημαντικά προβλήματα στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ όλους σας για τη συνεισφορά σας στην σύνταξη της έκθεσης. Ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος. Πολύ λιγότερο από 45 λεπτά. Τόσο λίγα που μας ε, λείπουν κάποιοι από τους σκιώδεις. Μάικλ. Μιλάω για τον κύριο Ζω. που ζητά συγγνώμη διότι δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα θέλει να ευχαριστήσει και να συγχαρεί τον εισηγητή για το έργο του. Λέει ότι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ σκιωδών του εισηγητών και του εισηγητού ήταν πολύ καρποφόρα, χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Το σχέδιο εκθέσεως βελτιώθηκε σημαντικά όσον αφορά τον ορισμό των ιδιαιτεροτήτων κάθε οργανισμού κυρίως. Το κείμενο επακριβώς καθορίζει τους διάφορους ρόλους και τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που πρέπει να εγγυάται την ειρήνη και ασφάλεια των πολιτών της επικράτειάς της και όσον αφορά τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ. Επίσης εντοπίζει βασικούς τομείς συνεργασίας συμπεριλαμβανομένη στρατιωτικής κινητικότητας, κάτι που συζητήσαμε το πρωί και σωστά υπογραμμίζει ότι η κίνδυνη επικάλυψης ή ανταγωνισμού είναι πολύ μικρή και ότι οι συμπληρωματικότητε θα πρέπει να τονιστούν. Το κείμενο τονίζει επίσης την ανάγκη συγκεκριμένης εφαρμογής των προτάσεων που υιοθετήθηκαν από τα δύο θεσμικά όργανα. Ο κ. Νταζόν ελπίζει ότι το σχέδιο εκθέσεως θα υιοθετηθεί με μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή αφετ αύριο το πρωί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Δεν έχουμε τον εισηγητή του ΙΣΙΑΡ εδώ. Πάμε στην κυρία Βότμανς λοιπόν για την Άλντε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Πάσκου. Πολύ καλή δουλειά που έκανε. Σε ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, περίπου 30 τροπολογίες υπέβαλε η Άλντε, κάποιες τροπολογίες που αφορούν τη Ρωσία. Εκφράσαμε ανησυχίες για τη συμπεριφορά της Ρωσίας. Πιστεύει ότι η Άλντε είναι ότι είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να διατηρήσει το διάλογο με τη Ρωσία και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται κοινή στρατηγική προσέγγιση εναντί της Ρωσίας. Έχουμε και κάποιο σχέδιο στην Άλτη όσον αφορά τι νέε σχέσει με τη Ρωσία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα. Η αδίποτε επιθετικότητα τη Ρωσία, υβριδική ή συμβατική, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο όταν ε, επιτίθεται και εισβάλλει στις ανατολικές χώρες, ε, στην ανατολική πτέρυγά μας, πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι συμπεριφορές. Η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ πρέπει να ισχυθεί όχι μόνο στην αριστερή πτέρυγα, αλλά και στην νότια πτέρυγα. Η Άλτα εξέφρασε επίσης τις συνέπειες που έχει το Brexit για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. 80% των αμυντικών δαπανών ε, του ΝΑΤΟ θα είναι, ε, δεν θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit. Τρεις από, από τα τέσσερα συντάγματα στην, Ανατολική Πτέρυγα θα ανήκει σε χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ευπρόσδεκτες οι δεσμευτικές ε, δηλώσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την ΠΕΣΚΟ για τη διάθεση χρημάτων για την άμυνα. Όσον αφορά την ΠΕΣΚΟ, η ΠΕΣΚΟ είναι εποφελής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον ΝΑΤΟ. Ε, αυτό πρέπει επανειλημμένα να τονίζεται. Τονίσαμε τη σημασία συμβατών δυνατοτήτων που διευκολύνουν ε, την ανάπτυξη των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Είναι ατυχές όταν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επιλέγουν μη, συμβατά, μη συμβατό εξοπλισμό, όπως η απόσταση της Τουρκίας να αγοράσει ρωσικούς ε, πυράβλους που δεν είναι συμβατή με τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ. Σχετικά με αυτό, αλλά και πιο γενικά, επίσης ζητούμε να γίνει διάλογος στον οποίο θα ηγεί το ΝΑΤΟ για να μειωθούν οι εντάσεις μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ, παραδείγματος χάρη μεταξύ ΙΠΑ ε, και Τουρκίας. Υπογραμμίσαμε επίσης ότι σε οποιαδήποτε επιχείρηση στα πλαίσια της διαχείρισης παράτυπης μετανάστευσης, καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα των ετούντων άσυλων και των μεταναστών θα πρέπει να γίνονται σεβαστά Είμαστε στην Ευρώπη και πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των μεταναστών. Επίση, υπάρχουν τεράστιε ευκαιρίε για συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση για, τους κυβερνα, για τι κυβερναπηλέ. Και προτείναμε διαγραφή παραγράφου που έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερα εξοπλισμένη για θέματα εσωτερική ασφάλεια και το ΝΑΤΟ καλύτερα για εξωτερική άμυνα. Αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό. Πολλέ από τι τροπολογίε μα ελήφθησαν υπόψη συμβαστικέ τροπολογίε και Άλτε θα υποστηρίξει όλες τι συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ και α προχωρήσουμε λοιπόν μέσα σε αυτή την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάιτμανς. Και τώρα ο κύριος Κουζούν Πεμρούι. Εμείς ε, έχουμε ξαναπεί ότι θα παρουσιάσουμε μία έκθεση μειοψηφίας δεν συμφωνούμε με τα όσα λένε οι περισσότερες ομάδες, ε, ούτε και ο Σπάσκου σε ό,τι αφορά την, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να υπάρχει και θα πρέπει να χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει, ε, τις του για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν αυτή την αμοιοψηφική έκθεση. Ευχαριστώ. κύριος Μεζέρικ. Σύντομος θα είμαι. Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Υπήρξε ουσιαστική βελτίωση του αρχικού κειμένου. Τώρα λαμβάνουμε υπόψη μας ε, περισσότερο τις ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια κενά Προσπαθούμε να ορίσουμε πιο καλά την έννοια, τη δύσκολη έννοια της συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών οργανισμών και τις ε, συμπληρωματικότητές τους. Πάντα αναφερόμαστε στην ε, συμπληρωματικότητα, συχνά ως σλόγγαν. Μερικές φορές όμως δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε. Ίσως είναι δύσκολη η απέτηση και είναι δύσκολο να το καθορίσει αυτό η έκθεσή μας, αλλά η ανησυχία μας είναι παλιά. Έχουμε πρόβλημα με τη χρηματοδότηση. Πιστεύουμε ότι για να βελτιώσουμε τη, ε, στις δυνατότητες θα πρέπει να ενισχύσουμε την ΠΕΣΚΟ. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ξοδεύουμε ενωσιακό χρήμα ε, για την στρατιωτική έρευνα, η ανάπτυξη. Αυτό είναι μεγάλη μας ανησυχία και δεν έχει διασκεδαστεί. Υπάρχει παραμένει λοιπόν. Και όπως αναφέρθηκε επίσης από τους συναδέλφους, δεν είμαστε πεπισμένοι ότι οι μη συμβατικές ρωσικές απειλές αφορμό την, την Ανατολική Ευρώπη. Αν πάρετε το Brexit, ε, το χακάρισμα της, του Υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας, το θέμα δεν είναι η αντιπαράθεση Ανατολής-Δύσης. Δηλαδή η Δύση ε, θα πρέπει να δούμε μάλλον ε, πώς θα βρούμε την αλληλεγγύη για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες και θα δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Κλείνουμε λοιπόν εδώ τις παρουσιάσεις των σκιωδών ομιλητών. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να μιλήσει. Επομένως, ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Πάσκου για να ολοκληρωθεί εδώ η συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά για τα σχόλιά σας, για την υποστήριξή σας. Όλες οι απόψεις είναι σημαντικές. Δεν θέλουμε για της βίας να πείσουμε τους άλλους ότι έχουμε τη σωστή άποψη ούτε κατά ανάγκη να καταπιούμε στις τι δικέ του απόψει. Θα πρέπει τουλάχιστον να ξέρουμε γιατί κάποιες θέσεις υιοθετούνται. Δηλαδή, να καταλάβουμε τουλάχιστον για ποιο λόγο κάποιοι υποβάλλουν ε, τροπολογίες ή έχουν επιφυλάξεις. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τη θέση τους. Επίσης, ε, ας αφήσουμε αυτή την επικοδομητική αμφισημία, ας πούμε, να βασιλέψει. Ένας υπέροχος όρος που επινοήθηκε από τους Βρετανούς. Ο, ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Μας σώζει μερικές φορές αυτή η επικοδομητική ασάφεια. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, έχουμε φτιάξει πολλές τέτοιες φράσεις εμεί οι Βρετανοί, η αγγλική γλώσσα. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, για την έκθεση και για τις τροπολογίε. Όπως και με την προηγούμενη έκθεση θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί στην ΑΦΕΤ και συνεχεία στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Αυτά. Ευχαριστώ. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η ετήσια έκθεση για την, τις αποστολές και επιχειρήσεις του 2017 της ΚΠΑ. Ο κύριος Ντίν, ο οποίος είναι διευθυντής της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, είναι εδώ και εκπροσωπεί το CPCC που είναι η μη στρατιωτική δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων. Uh, Κύριε Ντίν, καθίστε παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Είναι η δεύτερη ετήσια έκθεση για τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑ. Η πρόθεση ήταν να προκαλέσουμε και τον ε, στρατηγό που είναι επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους για αυτές τις αποστολές και επιχειρήσεις, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει. Ο κύριος Ντίν όμως θα μας παρουσιάσει τις επιτυχίες των πολιτικών αποστολών πέρυσι. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, αλλά θέλουμε να ακούσουμε ειλικρινή λόγια από εσά για τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν αυτές οι αποστολές και επιχειρήσεις και πώς βλέπετε το μέλλον αυτών των αποστολών. Τέλος, η CPCC, της οποίας είστε επικεφαλής, ε, συνδέεται στενά με το MPCC, ε, που είναι το στρατιωτικό σκέλος, ούτως ώστε να υπάρχει ε, η μέχρι δυνατή συνέργεια και συντονισμός το στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους. Και το MPCC και το JSCC θα αναθεωρηθούν φέτος από το Συμβούλιο. Πώς κρίνεται την λειτουργία του JSCC, που ενδιαφέρει φυσικά το CPCC, ε, έχουμε ένα καρό ακρονίμια δυστυχώς. Πολύ ωραία. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ντίν για να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Είναι πάντα χαρά για μένα να έρχομαι στην Επιτροπή σας και να μοιράζομαι μαζί σας και τα καλά και κακά μαντάτα και τις προκλήσεις. Όπως ξέρετε και από το παρελθόν, ε, θα σας εξηγήσω και τι πάει καλά και ποιες είναι οι προκλήσεις. Έχουμε περίπου 2.000 ε, άτομα στις 10 αποστολές σε τρεις υπήρους. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Ε, αρκετά σημαντικός μηχανισμός. Οι αποστολές μας γενικά τα πάνε καλά, θεωρώ είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε στην εργαλειοθήκη μας. Και δεν είναι ούτε καλύτερες ούτε χειρότερες από τις άλλες δυνατότητες που χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε κυρίως τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων των χωρών που μας χρειάζονται. Εγώ λέω ότι οι αποστολές είναι ένα πόδι ε, μιας καρέκλας με τρία πόδια. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα πολιτική οικονομική ασφάλεια. Και εμείς προσπαθούμε ακριβώς να είμαστε η ασφάλεια. Εάν όμως δεν υπάρχουν τα τρία σκέλη σε αυτό το σκαμνί, πέφτει όποιος πάει να κάτσει. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη. Είναι σημαντικό και αυτό για να δούμε δηλαδή πώς αντασσόμεθα στην γενικότερη ενωσιακή προσπάθεια. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε με ολιστικό τρόπο. Οι αποστολές μας δεν πρέπει να δρούν απομονωμένα από τα άλλα ενωσιακά ε, όργανα ή τις ε, άλλες παρεμβάσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ της Αφρικανικής Ένωσης. Από το 2004-2005 έχουμε ξεκινήσει αυτές τις αποστολές. Είμαστε λοιπόν σε πρώτη φάση. Θα μιλήσω και για τις στρατιωτικές και για τις μη στρατιωτικές. Νομίζω ότι ένα από τα πλεονεκτήματά μας δεν είναι μόνο οι λεπτομέρειες του τι κάνουμε. Γιατί έχουμε μία ετήσια έκθεση που αποφασίσαμε να αρχίσουμε να εκδίδουμε γιατί δεν πουλάμε αρκετά τις επιτυχίες μας στα κράτη-μέλη, στην κοινή γνώμη για να καταδείξουμε γιατί είναι σημαντική η δουλειά που κάνουμε. Αλλά η σημαντική πλευρά και αυτό που μας κάνει διαφορετικούς είναι ότι είμαστε πολύ ορατοί. Βλέπουν την ευρωπαϊκή σημαία, βλέπουν τις εθνικές σημαίες, βλέπουν τους στρατιώτες, τους αστυνομικούς, βλέπουν τι κάνουν. Είναι δηλαδή πολύ ορατή η παρουσία μας. Ιδιαίτερα εκεί που είμαστε πολύ άριθμοι, όπως στο Αφγανιστάν αλλά και στο Κωσυφοπαίδιο. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί πολλέ φορέ τα εργαλεία μα, παρά το ότι είναι σημαντικά και παρά το ότι δαπανούμε πολλά, δεν φαίνονται. Δεν φαινόμαστε επί Άρα, ίσω η Ένωση δεν λαμβάνει την αναγνώριση που της αρμόζει. Ότι η παρουσία μα δηλαδή παίζει ρόλο, αλλάζει την κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι είμαι υπόλογο και στα κράτη-μέλη φυσικά αλλά και έμεσα στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για τη στήριξη και τις κατευθυντήρες γραμμές που μου δώσατε. Γιατί κοστίζουμε. Κοστίζουμε γύρω στα 260 εκατομμύρια. Δεν είναι πενταροδεκάρες. Πρέπει λοιπόν οι επικεφαλείς των αποστολών να αξιοποιούν σωστά αυτούς τους πόρους. Να μην είμαστε απλώς πολιτική παρουσία. Πρέπει η παρουσία μας να αλλάζει τα πράγματα. Και θεωρώ ότι θέλουμε όντω και εγώ και το προσωπικό μας επιτόπου να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θέλουμε απλώς να είμαστε Κίνα για να δείχνουμε ότι είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να αποκτήσουν οι κάτοικοι των χωρών αυτών πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη χωρίς νεποτισμό και πολιτικές παρεμβάσει. Θέλουμε οι δυνάμει ασφαλείας των χωρών αυτών να είναι τμήμα τη λύση και όχι του προβλήματο. Γι' αυτό πολλέ από τι αποστολέ μα στο παρελθόν και ίσως λιγότερο τώρα έχουν συγκεντρωθεί στην πλευρά της αστυνόμευσης. Η αστυνομία είναι το πρώτο σημείο επαφής που έχει ο πληθυσμός με τις αρχές και στο παρελθόν ήταν τμήμα του προβλήματος. Είναι σωστό να αντιμετωπίζονται σωστά οι πολίτες από την αστυνομία και να έχουμε υπόψη τα θεμελιώδη όταν προσπαθούμε να αναπτύξουμε υπηρεσίες. Πρέπει να προωθήσουμε τους θεσμούς του κράτους δικαίου. Να είναι πραγματικοί θεσμοί του κράτους δικαίου. Να μην είναι πολιτικό όργανο στα χέρια οποιασδήποτε κυβέρνησης. Πρέπει να τα έχουμε υπόψη αυτά. Και πάντα τα έχουμε υπόψη αυτά. Είναι σημαντικό καθήκον και πρόκληση για να αλλάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, οι αποστολές μας στην αρχή ήταν αποστολές αστυνόμευσης. Και πρόσφατα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, προσπαθούμε να δούμε τη σχέση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Άρα ασχολούμεθα περισσότερο με τα θέματα μετανάστευσης. Γιατί η τρομοκρατία στους δρόμους μας έχει να κάνει με την κατάσταση αυτή. Στόχος μας είναι λοιπόν να προστατεύσουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες. Εγώ είμαι πρώην αστυνομικό και θεωρώ ότι η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από την αντιμετώπιση. Αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα στην πηγή και σε μερικέ από τι χώρε που δρούμε, δυστυχώ, αλλά όντω, είναι η πηγή μερικών από τι επιθέσει που αντιμετωπίσαμε στις δικές μας χώρες. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε διοργανικέ αντιζηλίες ή διαδικαστικές ε, διχογνωμίες να εμποδίσουν τη συνεργασία. Πρέπει να δρούμε όπως διακηρύσουμε. Όταν πηγαίνουμε σε αυτές τις χώρες, τους λέμε γιατί χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση. Γιατί οι δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να συνεργάζονται καλύτερα. Να καθορίσουν τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες και να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Άρα λογικό είναι ότι και εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. και όλες τις εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας που χρηματοδοτεί ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος. Και αυτό που κάνουμε και εξωτερικά. Έτσι θα κερδίσουμε όλοι. Αν βοηθήσουμε τους πολίτες μας, δηλαδή να τους προστατεύσουμε, να εξασφαλίσουμε τα σύνορά μας, να κάνουμε τις χώρες μας πιο ασφαλείς και αν παράλληλα βοηθήσουμε να αναπτυχθούν στις χώρες που δρούμε ανάλογες δυνατότητε, τότε θα επιτύχουμε κάτι ουσιώδες. Είναι μια σωστή φιλοδοξία. Σωστά πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θέλουν σε στρατηγικό επίπεδο να είναι ιδιαίτερα στοχευμένες αυτές οι αποστολές. Είναι σημαντικό. Γιατί τα κράτη-μέλη καταλαβαίνουν καλύτερα το στρατηγικό επίπεδο από το λειτουργικό τακτικό επίπεδο, αλλά το τακτικό επηρεάζει περισσότερο την κατάσταση. Εργαζόμαστε σε χώρες που είναι ακόμη σε συνθήκες ε, σύραξης ή μόλις έχουν βγει από αυτές και όπου τα καθεστώτα είναι πολύ αυταρχικά ή και δικτατορικά. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αν ελέγξεις σε αυτό το επίπεδο την κατάσταση, τότε και οι φυστάμενοι τους θα συμμορφωθούν. Πρέπει λοιπόν εφιώς να δούμε πώς θα προσανατολίσουμε τις προσπάθειές μας. Αναπτύσσουμε λοιπόν νομοθεσία, προσπαθούμε να καθορίσουμε τις ευθύνε και τις αρμοδιότητες των διαφόρων, των διαφόρων δυνάμεων ασφαλείας, της εθνικής φρουράς ή της αστυνομίας. Δεν συνεργαζόμαστε απευθείας με τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά όταν προσπαθεί να καθορίσει το επίπεδο ασφαλεία, ε, πρέπει να συνεργαστεί και με τι ενόπλε δυνάμει, έστω και εμέσα. <clears throat> και καταλάβαμε ότι δεν αρκεί η μεταρρύθμιση ενό κρίκου τη αλυσίδα. Δεν ε, παίζει μεγάλο ρόλο το να έχει καλή αστυνομία εάν δεν έχεις ε, καλό δικαστικό σώμα ή σωστά σωστά λειτουργών σοφρονιστικό σύστημα. Άρα πρέπει να υπάρχει και σωστή πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Πρέπει είτε οι πολίτες που έχουν διαπράξει αδικήματα ή αυτοί που, έχουν, που είναι θύματα πρέπει να έχουν σωστή πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε σωστή δικαιοσύνη. Και όταν κάποιος δικάζεται πρέπει να αντιμετωπίζεται δίκαια με βάση τους κανόνες που θεωρούμε ότι πρέπει να ισχύουν. Είμαι συνταξιοδοτημένος ε, αστυνομικός από τη Βόρεια Ιρλανδία Άρα ξέρω διαφορετικές ε, μεθόδους αστυνόμευσης, θα το πω έτσι. Τα τελευταία 11 χρόνια έχω ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Αλλά αυτό που θυμάμαι πάντα ήταν ότι υπήρχε τρομερή εξάρτηση από τις ε, ομολογίες. Οι ομολογίες βέβαια είναι καλό εάν έχουν ε, αποκτηθεί δικαίως και νομοτύπως. Αλλά αυτό που με εκπλήσει είναι ότι κατά τη δικαστική διαδικασία υπάρχει υπερβολική εξάρτηση από τις ομολογίες. Αυτό ενθαρρύνει την προσπάθεια απόσπασης ομολογιών. Το βασικό λοιπόν είναι να ισχύει πάντα το κράτος δικαίου, ανεξάρτητα αν κάποιος είναι θύμα ή θήτης. Όπως, είπα, έχουμε αποστολές σε τρεις υπήρους. Στην έκθεση θα βρείτε λεπτομέρειες. Εγώ θα είμαι συνοπτικός. Έχουμε στην Ευρώπη αποστολή στη Γεωργία, όπου ανησυχώ. Ξέρω ότι πήγατε πρόσφατα, γιατί ενδιαφέρομαι να μάθω τι έγινε εκεί, στο Κοσφοπέδιο και την Ουκρανία. Η αποστολή στη Γεωργία είναι από τον Αύγουστο του 2008 από τις παλιότερες και από τις πιο επιτυχημένες. Και το λέω ειλικρινά αυτό σε βάθος χρόνου. Δεν είναι εύκολη η αποστολή. Αλλά οι αποστολές επιτήρησης είναι πάντα πιο εύκολες από τις αποστολές μεταρρύθμισης. Γιατί και οι Ρώσοι αναγνωρίζουν, έστω και αν δεν λένε ότι εκτιμούν την ε, παρουσία μας, γιατί δυσχεραίνει τις προσπάθειες ε, προπαγάνδας και ψευδών ε, δηλώσεων και ειδήσεων. Η αποστολή μας λοιπόν έχει επιτύχει πολλά και υποστηρίζεται από τα κράτη-μέλη. Πολλά από τα κράτη-μέλη συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή. Είμαστε σε 23-24 τώρα στα χώρες. Κάποτε ήταν όλες οι χώρες. Γιατί πάντα μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι το επαρκές προσωπικό για την Ουκρανία που είναι πρόσφατη αποστολή. Ξεκίνησε χωρίς την καλύτερη εντολή. Μόνο στρατηγικές συμβουλές δίναμε σε υπουργικό επίπεδο και έπρεπε να δώσουμε πολλές συμβουλές σε πολλές οργανώσεις κυβερνητικές, μη κυβερνητικές και δεν επηρεάζαμε τα πράγματα. Τώρα η διεύρυνση για να έχουμε και πέντε επιχειρησιακές γραμμές για διερεύνηση εγκλημάτων, ε, δημόσια, τάξη και άλλες έρευνες, όλα αυτά είναι σημαντικά και την τοπική αστυνόμευση. Όλα αυτά μας έχουν δώσει πολύ περισσότερη και ορατότητα αλλά και δυνατότητα επίδρασης. Είμαστε σε τρία όμπλα στο Λβίβ, το Χάρκιβ και πρόσφατα και στην Οδυσσό. Το Φεβρουάριο ανοίξαμε γραφείο. Και είναι γενικώ ε, αποδεκτή. Αλλά οι προκλήσεις είναι βέβαια συλλογικέ. Κοσμοπέδια. Ε, περνάω ξάριμπνες νύχτες για αυτή την αποστολή. Είναι περίπλοκη. Γιατί έχει εκτελεστική εντολή που είναι να υπάρξει μεταρρύθμιση της αστυνομίας και των τελωνίων. Αυτά πήγε καλά. Αλλά η μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος είναι πολύ πιο δυσχερή. Εκεί γίνονται πολλές παρεμβάσεις. Είναι μικρή περιοχή. Και πολλοί γνωρίζουν πολλούς. Οι πάντες γνωρίζουν τους πάντες. Έχουμε επιτύχει πολλά. Αλλά είναι πολιτικό παιχνίδι. Τώρα είμαστε δέκατο χρονό, αναλάβαμε από την UNMEC, την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών. Το καλοκαίρι θα αρχίσουμε να μειώνουμε ή να βελτιστοποιούμε, όπως θέλετε πέστε το, από 800 500. Η εντολή θα είναι πολύ πιο επικεντρωμένη στις συμβουλές και λιγότερο σε εκτελεστική παρέμβαση. Θα διατηρήσουμε όμως την εκτελεστική εντολή γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε την αστυνόμευση και την προστασία των συνόρων. Έχουμε και εκτελεστικό ρόλο, άρα πρέπει να έχουμε τους ε, ανάλογους πόρους, αλλά και για τα ειδικά δικαστήρια, που θα ακούσουν, ε, θα, εκεί θα εκδικαστούν υποθέσεις που μπορεί να προκύψουν μετά την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2011. Μόλις προσλάβαμε ένα νέο εισαγγελέα που θα ασχοληθεί με αυτέ τι ενδεχόμενε δικαστικές υποθέσεις, τι ενδεχομένε διώξει. Η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας πολλοί μπορούν να θεωρούν ότι προωθεί κυρίω περιορισμένου χρόνου ε, αποστολές, αλλά οι περισσότερε βαστάνε τουλάχιστον 10 χρόνια. Έχουμε ένα ρόλο βεβαίω να παίξουμε. και βεβαίως ε, η αποτελεσματικότητα των αποστολών μας εξαρτάται από την πολιτική βούληση των ε, χωρών όπου εργαζόμεθα για να αναλάβουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και τη δυνατότητα απορρόφησης ε, αυτών που δίνουμε από τα κράτη-μέλη, από τα κράτη όπου εργαζόμεθα. Δεν έχει καμία έννοια να στείλουμε 100 συμβούλους να συμβουλεύουν 5 άτομα. γιατί ξέρετε ορισμένες φορές δεν είναι η έλλειψη συμβούλων, διεθνών συμβούλων από αυτές τις χώρες που, σε αυτές τις χώρες που λείπει, αλλά αντίθετα υπάρχει πληθώρα. Ορισμένες φορές όμως πρέπει να συντονιζόμαστε και καλύτερα και με τους άλλους φορεί που δίνουν συμβουλέ. Γιατί αν υπάρχουν διχογνωμίες μεταξύ Ένωση, για παράδειγμα, και Νομών Εθνών, τότε αμέσω θα τι αντιληφθούν ε, οι επιτόπου και θα τι αξιοποιήσουν. Πολλέ φορές στέλνουμε υπερβολικά πολλά άτομα για να ασχοληθούν με τον ίδιο τομέα, για να κάνουν μεταρρυθμίσεις και πιέζουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτό είναι πρόκληση. Το Κοσμοπέδιο είναι πιο επιτυχημένο παρόλα αυτά. Πιο επιτυχία, πιο επιτυχία παρά αποτυχία. Μίλησα για τη Γεωργία και για την Ουκρανία. Στην Αφρική έχουμε τη Σομαλία ξεκινήσαμε τη νέα επιχείρηση Νέστορ. Βασιδόζόμαστε βεβαίως και ως ε, εφεδρικό γραφείο στην ε, Κένια, στον Αερόμπι, αλλά κυρίως είμαστε στο, στην περιοχή Σομάλι Λάν, στο Μογκαντίσου. Έχουμε αυτήν την ε, επιχείρηση ασφάλειας των συνόρων, έχουμε το Amazon. Θα μειωθεί από ό,τι φαίνεται η αφρικανική παρουσία. Αυτό θα δημιουργήσει κενά σε ολόκληρη τη Σομαλία, άρα πρόβλημα. Όμως ε, εδώ έχουμε ανεπάρκεια. Έχουμε το 50% του προσωπικού που θα θέλαμε. Άρα πώς να επιτύχεις τους στόχους με τους ε, μισούς πόρους. Τα κράτη-μέλη ψηφίζουν ε, με τα πόδια τους εάν θεωρούν ότι κάποιος τομέας της εξωτερικής πολιτικής δεν έχει έννοια. Δεν θέλουν να πληρώσουν το κόστος εάν δεν έχει αποτελέσματα. Αλλά αυτό είναι πρόκληση. Κάθε οργάνωση, για κάθε αποστολή ε, μπορεί να τα καταφέρει μόνο στο βαθμό που έχει το κατάλληλο προσωπικό. Αλλά γενικά παρά τις ελλείψεις προσωπικού αυτοί που στέλνονται είναι πολύ καλοί, πολύ κατάλληλοι. Αυτοί που πάνε στις αποστολές είναι άτομα τα οποία είναι ενεργά επαγγελματικά, δεν είναι συνταξιούχοι που έχουν ξεχάσει τι πρέπει να κάνουν. Οι αστυνομικοί από οποιαδήποτε χώρα βεβαίως βασίζονται και στη στήριξη που έχουν από τα Υπουργεία τους, ε, τα σώματά τους, τις κυβερνήσεις τους και αυτό τους δίνει ένα πλεονέκτημα. Πολύ διαφορετικό από το να είσαι απλώς κάποιος ε, ανεξάρτητος σύμβουλος Βεβαίως κάποιοι ανεξάρτητοι σύμβουλοι από ιδιωτικούς οργανισμούς μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν. Αλλά εμείς έχουμε αυτή την επιπλέον, το επιπλέον κύρος, γιατί μιλάμε ως Ευρώπη. Δεν μιλάμε απλώς ως ε, διαχειριστές ενός προγράμματος, αλλά η Σομαλία είναι πρόβλημα. Καλά τα πάει η αποστολή μας στο Μογκαντήσου. Καλά πάει και η Ατλάντα, η Unifor, ε, η θαλάσσια. Κοιτάξτε, η πειρατεία δεν πρόκειται να σταματήσει, γιατί είναι πολύ επικερδής. Πολλοί από αυτού ε, είναι βεβαίω εγκληματίε, μπορείτε να σου πείτε ό,τι θέλετε. Και ξέρετε, αν τους κόψουμε μία δυνατότητα να επιτίθενται σε πλοία, ε, θα περάσουν σε άλλες δραστηριότητε. Μπορεί να κάνουν διακίνηση ατόμων, αποσπούν χρήματα δηλαδή από τα θύματα. Γι' αυτό πρέπει να αυξηθούν οι τοπικές δυνατότητες αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων. Στο Σαχέλ, Μάλι και Νιζέρ, καλές αποστολές. Στο Νιζέρ γίνεται πολύ καλή δουλειά, παρατηρούμε και αυξάνουμε τις δυνατότητες της κυβέρνησης εκεί για να αντιμετωπίσει την παράτυπη μετανάστευση κάπως καλύτερα και το έχω συνδέσει καλά με την αποστολή μας στη Λιβύη, κυρίως στη Βόρεια Λιβύη, ούτω ώστε αυτές οι δύο χώρες και το Μαλί και η Αλγερία να συνεργαστούν για καλύτερο έλεγχο των συνόρων τους και παρακολούθηση της δραστηριότητα. Οι αποστολές Μάλι Νίζερ είναι πολύ σημαντικές. Στον Παμάκο είναι το κέντρο. Εξετάζουμε και τις χώρες G5, Τσάντ, Μαυρετανία και Μπουρκίνα Φάσο δηλαδή, για να διασφαλίσουμε την ε, συνεργασία μεταξύ αυτών των χωρών στον πολιτικό και στρατιωτικό τομέα για να ελέγχονται τα σύνορα να είναι πολύ πιο στεναρά για να αντιμετωπιστεί και η τρομοκρατία και η μετανάστευση και η λαθρέα διακίνηση ατόμων και αγαθών. Η Λιβύη για λόγους που κατανοείται είναι δύσκολη περίπτωση. Αλλά χαιρόμαστε και αρκετά υπερήφανοι είμαστε, αλλά η παρουσία μας στη Λιβύη μαζί με την παρουσία κρατών μελών Τριπλασιάστηκε η παρουσία μας λοιπόν. Δεν θέλουμε όμως να είμαστε οι μόνοι παρόντες. Η επιτυχία μας θα είναι εάν μειώσουμε την παρουσία μας, να αντικατασταθεί αυτή η παρουσία από τις τοπικές αρχές. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση. Θα τελειώσω για τρία λεπτά, Πρόεδρε. Ξέρετε τι έχει γίνει στη Μέση Ανατολή τι τελευταίε μία-δύο μέρε, οπότε καταλαβαίνετε τι προκλήσει αντιμετωπίζουμε. Η αποστολή μα στη Ραμάλα. Έχουμε συναδέλφου στη Ιερουσαλήμ. Όλοι αυτοί τα έχουν πάει πολύ καλά. Η μεταρρύθμιση τη ε, Παλαιστινιακή αστυνομία τα πάει πολύ καλά. Αλλά μόνο στην Δυτική Όχθη. Δεν καλύπτει την Γάζα. Η αποστολή μα στη Ράφα ε, είναι ανενεργία το 2007. Ήμουν στην Ράφα πρόσφατα, ελπίζοντα να βοηθήσω να υπάρξει συμφιλίωση μεταξύ Χαμάς και Φατά, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις θα δυσχεράνουν πολύ αυτή την εξέλιξη. Και τα κράτη-μέλη καταλαβαίνουν ότι δεν θέλουμε το προσωπικό μας να κινδυνεύει, θέλουμε να μειώσουμε τους κινδύνους από την παρουσία μας, για το προσωπικό μας δηλαδή. Η Ράφα λοιπόν θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολη, αλλά είναι παρούσα παρούσα ας πούμε ως δήλωση πρόθεσης. Και Ιράκ, η πρώτη εξαμηνία έκθεση της αποστολής ε, υποβλήθηκε χθες στην Πολιτική Επιτροπή Ασφάλειας. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι με το πώς προχωράει αυτή η κατάσταση. Είναι ακόμη μικρή, 36 άτομα. Ε, εργάζονται με το γραφείο του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας για να καθοριστούν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες Στο Ιράκ κυρίως ασχολούμεθα με στρατιωτικά θέματα για κατανοητούς λόγους, αλλά δεν θέλουμε να συνεχιστεί έτσι. Από τους ε, υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους με τους οποίους συνομιλώ, θεωρώ ότι καταλαβαίνουν τη σημασία του να υπάρξει μια πιο φυσιολογική, πιο δημοκρατική κοινωνία. Να υπάρχει ε, σωστή διακυβέρνηση και να εκτελούνται οι πολιτικές διαδικασίες από πολιτικές αρχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κάθε σεβασμό για τις στρατιωτικές αρχές που εφαρμόζουν τις πολιτικές διαδικασίες και πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος γι' αυτό. Αλλά θα μιλήσω για το στρατιωτικό τώρα θέμα. Ο στρατηγός Σπέκανεν δεν είναι εδώ, αλλά θα το αντικαταστήσω. Εργαζόμαστε από τις Βρυξέλλες γι' αυτό. Η, η επιτυχία εξαρτάται από το να δράσει το σωστό άτομο στη σωστή στιγμή και στη σωστή ε, διάσταση και στο σωστό ε, σημείο. Και δεν έχει σημασία αν είναι στρατιωτικός ή όχι. Πρέπει βεβαίως ε, να υπάρχει συνεργασία. Εάν πρέπει να υπάρχει και πολιτική και στρατιωτική λύση, το σημαντικό δεν είναι ποιο είναι πιο σημαντικό. Ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν δικογνωμίε από αυτού. Το βασικό είναι να δράσουμε με αυτέ τι τέσσερι σωστέ παραμέτρου. Υπάρχει λοιπόν ο στρατιωτικό σχεδιασμό που κάνει κάτι παράλληλο σε αυτό που κάνουμε εμεί στον πολιτικό σχεδιασμό, από πλευρά αποτελεσμάτων, πλευρά υποβολή εκθέσεων, λογοδοσία ούτως ώστε να δρούμε σε συνεργασία και με τους άλλους, να καταλάβουμε ότι είναι τμήμα της ευρωπαϊκής προσπάθειας για να εκπροσωπήσει όλες τις κράτη της Ένωσης, τα κράτη της Ένωσης, για να δώσουμε το παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να παίζουμε αυτό το ρόλο. Είναι καλό λοιπόν να υπάρχει συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής δράσης και μάλιστα να βρούμε σωστά επιτόπου. Στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν μεταξύ κοινέ αποστολέ. Υπάρχουν υπέρ και κατά, αλλά θα το εξετάσουμε. Πρέπει να δούμε πώς συνεργαζόμεθα. Και τα κράτη-μέλη και θεωρώ και το Κοινοβούλιο απαιτούν να υπάρχει περισσότερο συντονισμός η κύρια πρόκληση υπάρχουν διάφορες. Αλλά υπάρχουν ορισμένες που αφορούν όλες τις αποστολές. Πρώτα απ' όλα επαρκή πόροι. πολύ λίγες από τις αποστολές μας έχουν επαρκές προσωπικό. Και μιλάω προσεκτικά, αλλά πρέπει να, σας, να είμαι ειλικρινής εναντί σας. Και το καταλαβαίνω. Μερικά. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι. Αλλά για να παίξουμε το ρόλο μας, να αλλάξουμε την κατάσταση, πρέπει να έχουμε επαρκείς πόρους, επαρκές προσωπικό. Και μερικές από τις μικρότερες χώρες δεν έχουν ε, ίσως ε, αρκετούς εμπειρογνώμονες και χρειάζονται πολλούς από αυτούς στη χώρα τους. Χρειάζονται στις ίδιες τους τις χώρες. Στα Υπουργεία Εσωτερικών Δικαιοσύνης. Και είναι απρόθυμοι να στείλουν άτομα 3.000 χιλιόμετρα μακριά όταν, τους, όταν τα χρειάζονται. Αυτό θα συνεχίσει να είναι πρόβλημα. Ξέρω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξέρω ότι τα Υπουργεία Εξωτερικών προσπαθούν να ενθαρρύνουν τα άλλα Υπουργεία για να στείλουν τους σωστούς εμπειρογνώμονες. Γιατί οι σωστοί εμπειρογνώμονες θα έχουν αποτελέσματα. Βεβαίως, ένα άλλο πρόβλημα είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει το προσωπικό μας επιτόπου. Τα τελευταία δέκα χρόνια είχαμε τέσσερα θύματα. Μπορεί να μην φαίνονται πολλά, αλλά έχουν οικογένειες, έχουν φίλους. Και η ασφάλεια του προσωπικού μας ε, μας αφορά, μας απασχολεί και είναι ακριβή. Πρέπει λοιπόν ε, να δαπανηθούν σωστά, ίσως να έχουμε οικονομίες κλίμακα στο μέλλον. Αν συνεργαστούμε με τις στρατιωτικές αποστολές. Γιατί εργαζόμεθα συχνά με ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλεια για πολλού λόγου. Αναφερθήκαμε στη Λιβύη για παράδειγμα. Ούτε η Λιβύη, ούτε το Ιράκ, ούτε το Αφγανιστάν είναι ασφαλή, ε, ασφαλείς χώρες και γι' αυτό κλείσαμε την αποστολή μας ε, στο Αφγανιστάν πρόσφατα. Και το Μάλι γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια. Αλλά να πληρώσουμε και το ποσό που χρειάζεται γι' αυτό. Ο κίνδυνος επίσης είναι της ε, διαφθοράς, ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές οι προσπαθίε μας από τις τοπικές αρχές. Αλλά όλα αυτά είναι αναμενόμενα, γιατί αν ήταν εύκολη κατάσταση δεν χρειαζόταν η παρουσία μα. Ανησυχώ πως πολλές φορές ε, είναι πολύ άνετη η κατάσταση των αποστολών μας γιατί θα είμαι ειλικρινής. Κανείς δεν θέλει να μεταρρυθμιστεί. Πολλοί με τους οποίους συζητάμε που θα πρέπει να υπογράψουν τις μεταρρυθμίσεις δεν τις θέλουν. Γιατί πολλές φορές θα χάσουν ίδια η εξουσία. Αλλά φυσικά δεν είναι εύκολο όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις διαφθοράς έλλειψης πραγματικής ε, πολιτικής προσέγγισης και καμιά φορά λένε πολλά λόγια και δεν κάνουν τις μεταρρυθμίσεις σε κάποιες χώρες, διότι δεν έχουν στερνιστεί την αποστολή. Λοιπόν, συντομία, 2.000 άνθρωποι, 10 αποστολές, κάποιοι καλοί άνθρωποι, άντρες και γυναίκες. Είχαμε πέντε γυναίκες στον επικεφαλής αποστολών της 10. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ηγούμεθα στις, σαν παράδειγμα. Τώρα έχουμε τρεις γυναίκες που είναι επικεφαλής αποστολών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό όταν συζητούμε με άλλους πολιτισμούς και μιλάμε ισότητα φίλων, και ισοτιμία και δικαιοσύνη και διαφάνεια θα πρέπει, και βλέπουν μόνο το ένα να εκπροσωπείται στην άλλη πλευρά του τραπεζιού δεν είναι Σωστό. Το κάνουμε λοιπόν ότι... γιατί είναι σημαντικό να έχουμε τις γυναίκες. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι γυναίκες είναι καλοί άνθρωποι, αλλά θέλουμε να, είναι, να έχουμε σωστή ε, εκπροσώπηση των γυναικών. Γιατί έχει αντίκτυπο. Πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Κυρία Πρόεδρε, μακρηγόρησα ίσως. Με τα χαράς να δώσω ειλικρινείς απαντήσεις. Σε έξι μήνες ολοκληρώνω τη θητεία μου απόλαυσα τις ε, προκλήσεις που αντιμετώπισα στη θέση μου και πιστεύω στη ΚΕΠΑ δεν είναι το μόνο σημαντικό εργαλείο, αλλά είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και σε κάθε αποστολή που πηγαίνω προκαλώ τους συναδέλφους μου. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη τους λέω. Δεν είσαστε εδώ για τα λεφτά. Μπορείτε να κάνετε διαφορά. Αλλά αυτό συνεπάγεται ευθύνε. Και ευθύνη ε, συνεπάγεται λογοδοσία. Λοιπόν, και γι' αυτό Είμαι λογοδοτό στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη και ευχαριστώ την Επιτροπή σας και την Επιτροπή ΑΦΕΤ για τις ε, προκλήσεις που μου ανέθεσαν, αλλά υποστήριξα, έτυχα υποστήριξης, ε, μου δόθηκαν σωστές συμβουλές. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να παρουσιάσω αυτή την επισκόπηση. Ευχαριστούμε κύριε Ντίν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντίν, λέει πρόεδρος. Ήταν ε, τι να σας πω, τελικά περιγράψατε πλήρως ε, το έργο το οποίο ηγηθήκατε και στο οποίο έχετε εμπλακεί και το εκτιμά το έργο σας η Επιτροπή πραγματικά. Και πιστεύω ότι εκφράζω και του συναδέλφους λέγοντας αυτό. Καταρχάς να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ το λόγο, το συνάδελφο, που ήταν μαζί μου στη Γεωργία την περασμένη εβδομάδα, πέραν όλων Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντίν. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Λυπούμεθα που τελειώνετε το έργο σας έξι εβδομάδες και συνάδελφοί μου και εγώ σας ευχόμεθα ό,τι καλύτερο. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε δυνατότητα να παραμείνετε στην Ένωση αν το επιθυμείτε. Είναι εύκολο αυτό για ανθρώπους που κατοικείτε στο δικό, στο δικό σας τμήμα της νήσου. Θα δούμε τι θα συμβεί τελικά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Πράγματι υπάρχουν κάποια ζητήματα πέρα από την περιγραφή των πεπραγμένων του περασμένου έτους και την ποσοτικοποίηση των επιτευγμάτων μας και πού βρισκόμαστε. Κάτω το παρελθόν, με άλλες εκθέσεις, ήδη ακούσαμε επικρίσεις. Σύμφωνα με αυτές, δεν θα έπρεπε μόνο να επιχειρηματολογούμε περιγραφικά ή ποσοτικά περί των επιτευγμάτων μας, αλλά να αναφερόμαστε και στους στόχους μας, τι θέλουμε να πετύχουμε. Βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών, μεγάλος στόχος αυτός Φερρυπίν. Ή αν είναι απομακρυσμένο το μέρος που δραστηριοποιηθούμε θα, ε, εάν έχουμε πετύχει κάτι σε σχέση με την έναρξη της αποστολής προς το τέλος της αποστολής. Και αυτή η αξιολόγηση ίσως να λείπει κάπως ε, από την παράθεση των διαφόρων αποστολών. Ίσως σε μελλοντικές εκθέσεις αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί. Και άλλο θέμα Αναφερθήκατε στους πόρους, κυρίως στους ανθρώπινους πόρους. Το πρόβλημα τόσο πολύ οικονομική πόρη, αλλά οι Σημειώσαμε σε πρώτες εκθέσεις ότι μόνο 75% των θέσεων στις πολιτικές αποστολές καλύπτονται και λυπούμεθα που ο κανονισμός προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα παρήχε καλύτερη προστασία και συνθήκες στο προσωπικό δεν ισχύει για προσωπικό που είναι στις αποστολές, που αποσχολείται από τι αποστολές, παρόλο που πληρώνονται από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό εμποδίζει την αποτελεσματικότητα των αποστολών και παροτείναμε τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι καλύπτονται οι θέσεις καταρχάς και μετά. Το ρώτημα είναι, γίνεται συζήτηση για την κάλυψη των θέσεων και αυτό το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί και να πούμε ότι εφαρμόζουμε τον κανονικό του περιπροσωπικού και σε αυτούς που συμμετέχουν σε αυτές τις αποστολές. Θα πρέπει να συζητηθεί αυτό, είναι απαραίτητο. Ίσως εσείς ε, πιέζετε, η ερώτηση είναι πιέζετε σχετικά με αυτό το θέμα και εσείς τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ Μάικλ. Χαβιέ. Ευχαριστώ. Μιλήσατε για το πρόβλημα των πόρων. Ε, εγώ δεν συμφωνώ ε, είναι πρόβλημα εντολής, βιώσιμη εντολή και συνέχεια ούτω ώστε να λειτουργήσει αυτή η εντολή. Να σας δώσω διάφορα παραδείγματα. Δεν μπορείτε να λέτε ότι η αποστολή μα στη Λιβύη είναι καλή όταν ο ευτέρο μας είναι ο Φαγέρα σαρά, ο οποίος ελέγχει το, το μέγαρό του στην Τρίπολη. Ε, και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Στο νότιο της Ευρώπης της Λιβύης, ξέρετε ότι υπήρχαν διάφορες πολιτοφυλακές και διάφορες ομάδες του Μισράτα. Και ξέρετε ότι διάφοροι εχμαλωτίστηκαν από αυτές τις πολιτοφυλακές. ο Χαλίφης Χάφτερ ε, ελέγχει τις ακτές. Υποτίθεται ότι είναι ακτές της ε, Λιβύης και όμως τις ελέγχουν ε, αλίτες. Πώς λέτε λοιπόν ότι έχουμε ε, συνεργασία με τον Ήγηρα. Ε, εσείς ε, μιλήσατε με τον Υπουργό που είναι έξινος άνθρωπος και ξέρετε για τι μιλάει. Ε, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αδύνατον όμως να συνεργαστούμε με, τον, ε, με την κυβέρνηση της, ε, ε, εκεί γιατί δεν ελέγχει τίποτα. Επομένως μιλάμε για σπατάλη, γιατί ο εταίρος μας δεν υφίσταται στην πραγματικότητα. θα πρέπει ε, επίσης να δείξουμε ρεαλισμό, όπως δείχνουμε στη Σομαλία, όπου ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι ε, που είναι παράνομο, η Σομάλιλαντ, με την οποία συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε γιατί είμαστε αναγκασμένοι. Ε, γιατί από την ακτή της Σομάλιλαντ ε, βγαίνουν διάφοροι πειρατές. Αν δεν έχουμε ένα πραγματικό εταίρο για να συνομιλήσουμε, δεν έχει κανένα νόημα Ε, γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι σχεδίες οι οποίες κινούνται ας πούμε προς κάθε κατεύθυνση. Γιατί να έχουμε τόσο μεγάλες αποστολές αν δεν παίζουν ρόλο. Να αναφέρω με παράδειγμα, Η γεωσυνογεωργία μας ήταν επιτυχημένη, ήταν θαυμάσια επιχείρηση. Αλλά ας πάμε τώρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ήμουν στην, στις εκπαιδεύσεις που κάνει η ΕΟΤΕΜ και είναι ντροπή, όχι για τους στρατιωτικούς που είναι εκεί, όχι για αυτούς που είναι εκεί, γιατί η πραγματικότητα τι είναι. Άμα δούμε ότι το έδαφος που γίνεται η εκπαίδευση είναι μια, ένα, ένα παρθένο δάσος. Όταν ε, η εκπαίδευση γίνεται χωρίς όπλα. Αυτό συμβαίνει. Και μετά έρχονται οι Ρώσοι και δίνουν όπλα και κάνουν αποτελεσματική εκπαίδευση. Και η επιχείρησή μας δεν εξυπηρετεί τίποτα. Παρά για να λέμε ωραίους λόγους ότι κάνουμε προσπάθεια στην κεντρική, κεντροαφρικανική δημοκρατία. Εάν ήμασταν κεντροαφρικανοί, μαύροι, θα βρίζαμε την ΕΟΤΕΜΕ όπως τη βρίζουν, που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μία αδύνατη εκπαίδευση έναντι της Σελέκα ή Αντιβαλάκα που αυτοί μπορούν να αγοράσουν όπλα. Είμαστε ιδιαίτερα υποκριτέ. Λέμε ότι τους εκπαιδεύουμε χωρίς όπλα για να πάνε να σκοτωθούν έναντι ληστών που έχουν όπλα και τα αγοράζουν πολύ φθηνά είναι τα υπόλοιπα από τον πόλεμο του Νταρφούρ από τους ε, αντάρτες Σανιουίτ. Μάλι. Έχω πάει επανειλημμένα. Και κάθε, κάθε φορά φεύγω όλο και πιο ανακτισμένος. Γιατί κάνουμε ακριβώς το ίδιο μετά από πέντε χρόνια εκπαίδευσης δεν έχουμε εκπαιδεύσει ούτε ένα λόγο 120 ανδρών, ούτε μία, ούτε ένα λόγο. Και ενώ προηγουμένω οι αντάρτες ήταν στο Κιδάλι και στο Τεσσαλί, τώρα είναι ε, έξω από το Μόκτη. Αυτό είναι σκάνδαλο. Γιατί όταν στείλαμε τους ε, χωροφύλακε του ΚΑΠ Μαλή, που ήταν καλά εκπαιδευμένοι, σταμάτησε να του πληρώνει η κυβέρνηση. Από τι θα ζούσαν λοιπόν έκλεβαν, έκλεβαν τους νομάδες Πέλ και τους νομάδες του Αρέγ από τον Τουαράγου και τον Χουμβαρί. Και τι θα κάνανε τότε αυτοί, εξεγέρθηκαν. Με τι, με τα όπλα που πήραν από ποιον, από το Αντσαρεντίν και από το Ιζάτα Γκάλι. Κατά συνέπεια, έχουμε μια τεράστια εξέγερση των Μπέλ εκεί που δεν υπήρχε προηγουμένω τίποτα. Και στην περιοχή Μενάκα, όπου υπήρχε ασφάλεια προηγουμένω από τι ομάδε του Αρέγ και του συμμάχου του κατά την Αντολαθώνα, επειδή είναι πολιτοφυλακές, τώρα είναι πολιτοφυλακές του Ασχράουι, που είναι τρομοκρατικές. Εάν μιλήσει λοιπόν ε, κανείς με αυτούς που δρούν επιτόπους, αν μιλήσει κανείς με τον πρώτο του Μπουρκίνα Φάσο, ε, Ροκ εάν μιλήσει κανείς με τους υπευθύνους, τους πραγματικά υπευθύνους στο Νιζέρ, καταλαβαίνει ότι η παρουσία μας δεν κάνει τίποτα αποτελεσματικό. Η Γαλλία το κάνει με την επιχείρηση Μπαγζόν και η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών. Η πολύ αποτελεσματική και αδυσόπιτη στρατιώτη του Τσάντ. Εγώ δεν λέω ότι είστε εσεί για όλα αυτά. Υπεύθυνη είναι η δική μα υποκρισία. Χωρί δυνατή εντολή. Χωρί αποτελεσματική παρακολούθηση. Χωρί ουσιώδη εκπαίδευση με όπλα. Γιατί οι εχθροί έχουν όπλα που σκοτώνουν. Του στέλνουμε να σκοτωθούν. Λόγω τη ε, υποκρισία μα Χρειαζόμαστε ουσιώδη εντολή, ουσιώδη παρακολούθηση και σε αυτή την περίπτωση και ουσιαστική χρηματοδότηση. Μόνο αν υπάρχουν τα δύο προηγούμενα. Άρα στην ουσία τον χρηματοδοτούμε κάτι το εντελώς ε, άσκοπο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ Χαβιέ. Σε αυτό το στάδιο δεν βλέπω να ζητάει κάποιος το λόγο άλλος και δράτω με τις ευκαιρίες να μιλήσω εγώ. Καταρχάς, όπως είπατε, είχαμε αποστολή στη Γεωργία της ΣΕΝΤΕ την περασμένη εβδομάδα και επισκεφθήκαμε την αποστολή από πλευρά Αυκασίας. Συνήθως πάμε στην Νότια Σετία. Και πήγαμε στο Ζιγδάτι και όπως είπατε είναι μια αποστολή που την έχουν υποδεχτεί οι ντόπιοι πάρα πολύ καλά, αλλά έχει και αποτελέσματα. εάν υπάρχουν ανησυχίες καταγγελίες, λειτουργεί η κόκκινη γραμμή, η γραμμή επικοινωνίας και αποκλιμακώνονται εντάσεις που αλλιώς θα είχαν κλιμακωθεί και είχαν δημιουργήσει και άλλα προβλήματα, όπως έχει συμβεί κατά το παρελθόν. Ο Χαβιέ το είπε. Είναι μία από τις αποστολές που πραγματικά είναι επιτυχής. Προφανώς θα παραταθεί τέλος αυτού του χρόνου για άλλα δύο χρόνια. Και αυτό που είπατε για το χρονοδιάγραμμα των αποστολών θα είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση η UMM, αυτή η αποστολή στη Γεωργία, να παραταθεί. Διότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Υπό δυσχερείς περιστάσεις. Κυρίως πρόσφατα και κυρίως στην περιοχή της Νότιας Οσετίας. Ένα-δύο άλλα σημεία που αναφέρατε. Αναφερθήκατε στην επικοινωνία. Πώς επικοινωνούμε με τους πολίτες μας η Γεωργία είναι άριστο παράδειγμα κατά πόσο πόσο φαίνεται στη Γεωργία η προσπάθεια που κατάβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γεωργία καλά τα πάει να παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Εμείς όμως εδώ στην επικοινωνία με τους πολίτες δεν τα πάμε τόσο καλά. Τι προβλέπετε ότι μπορεί να βελτιωθεί. Τι υποστήριξη χρειάζεστε για την επικοινωνία αυτή να είναι πιο αποτελεσματική η επαφή με τους πολίτες. Αναφερθήκατε στη Σομαλία. Αναφερθήκατε και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όπου η δραστηριότητα ξεφεύγει κάπως και επισέρχεται σε άλλες δραστηριότητες. Χρειάζεται ευελιξία, προσαρμοστικότητα όσον αφορά την εντολή για δράση. Μπορεί να παρασχεθεί μεγαλύτερη υποστήριξη και ευελιξία. Ή η παρέκκληση αυτή που διαπιστώνεται είναι η καλύτερη επιλογή. Για το θέμα της ισότητας των φίλων που αναφερθήκατε και ότι πάει καλά αυτό, χαίρομαι. Και άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο θέμα της τελέχωσης. Αν έχει την καλοσύνη να απαντήσετε. Α, και στον κύριο Γκάλερ δίνω το λόγο πάλι. Σωστά άκουσα ότι η αποστολή Γιούλεξ στο Κωσυφοπαίδιο ε, λίγη Η Γιούλεξ στο Ο όλεξ απάντησε εκτός μικροφώνου. Α, παρατάθηκε. Τότε τι άκουσα εγώ. Λοιπόν, διαγράψτε το από τα πρακτικά. Δεν έχω ερώτηση συμπληρωματική. Θα κάνουμε ότι δεν το είπατε καν αυτό, Μάικλ. Απάντηση. Για τον κύριο Γκάλερ. Όσον αφορά τις εκθέσεις, είναι η δεύτερη εκθέση που ετοιμάσαμε. Θέλουμε να ενημερώνουμε το κοινό. Θέλουμε να είναι περιεκτική, σύντομη, να περιγράφει το τι κάνουν οι αποστολές. το κοινό στις Βρυξέλλες δεν γνωρίζει καν την ΙΚΕΠΑ και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους μας είπαν πρέπει να μας πείτε τι κάνετε. Αυτό είναι καλό. Ίσως είναι ενηγματικά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κάτι μυστικιστικό. Αν ήξεραν ήξεραν τι κάνουμε ακριβώ ίσω σε δημοψηφίσματα ο κόσμο να ψήφισε διαφορετικά. Πρέπει να δείξουμε τι κάνουμε. Και ΚΕΠΑ είναι ένα από τα ορατά εργαλεία. Φορούμε στολέ, έχουμε σήματα κλπ. Είμαστε ορατοί. Και δαπανώνται πολλά εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι αξιέπαινα τα έργα που προωθούνται. Και δεν υπάρχει διεθνή αναγνώριση. Και πολύ συχνά εμεί πληρώνουμε, αλλά δεν έχουμε την αναγκαία θέση στο προσκήνιο και χρειάζεται να έχουμε μεγαλύτερη πρακτική παρουσία. Είναι κρίμα που οι πληθυσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξέρουν τι κάνουμε. Καλή φορά μας ξέρουν καλύτερα στις χώρες που δραστηριοποιούμεθα παρά στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 75% για, το, για τις θέσεις, περίπου 70-75% του προσωπικού έχουμε σε αποστολές. Κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν γύρω στο 80%. Το κενό είναι περίπου 20%. Όταν είσαι 70 με 80% σε τέτοιου είδους οργανισμούς θεωρείσαι πλήρως τελεχωμένος. Ποια είναι η αλήθεια όμως. Ενθαρρύνουμε, παρακαλούμε τα κράτη-μέλη. Σε κάθε εμφάνισή μου ζητήσαμε από την κυρία Μογκερίνη να το τονίζει αυτό. Μιλήσαμε σε, με ανθρώπους από τα Υπουργεία να τους ενθαρρύνουμε δεν μπορούμε να πιέσουμε τον κόσμο να έρχεται στις αποστολές μας. Στις πολιτικές αποστολές, το κάθε μέλος είναι θελοντές. Κάνουν αίτηση και υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτό είναι και πλεονέκτημα. Και οι άνθρωποι στη θέση μου λένε, χαμηλώνουμε τις προδιαγραφές μας για να έχουμε περισσότερο κόσμο. Καμιά φορά όμως δεν πρέπει να φέρουμε λάθος άνθρωπο με λάθος δεξιότητες, γιατί χάνουν όλοι έτσι. Δηλαδή έχουμε πλήρη στελέχωση αλλά δεν πετυχαίνουμε τα σωστά αποτελέσματα και στόχος μας είναι να κάνουμε τη διαφορά πετυχαίνοντας αποτελέσματα με ανθρώπους με τις σωστές δεξιότητες, σωστή θέση. Έχουμε αυτό το θέμα λοιπόν. Στο Σαχέλ είναι το θέμα της, ε, εκείνων που γνωρίζουν τα γαλλικά και μιλούν τα γαλλικά πρέπει να έχουμε προσωπικό που μιλεί τη γλώσσα, πρέπει όλα τα, μέλη της αποστολής να γνωρίζουν πολύ καλά τα γαλλικά, ίσως όχι. Χάνουμε μέλη της αποστολής που έρχονται σε επαφή με ανώτερα στελέχη στο Νίγηρα, στο Μαλί, στο Μπουρκίνο Φάσο, ίσως για πολλούς λόγους χάνουμε. Στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ χρησιμοποιούμε διερμηνείς και μεταφραστέ. Σω πρέπει να βρούμε πιο καινοτόμου τρόπου για να διορθώσουμε τα προβλήματα των πόρων. Να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα να μην αφήνουμε κάποιου ανθρώπου εκτό λόγω αυτού του προβλήματο. Είναι καλύτερα να μην έχουμε κάποιον στη θέση, κανένα στη θέση, διότι δεν μπορούμε να βρούμε γαλλόφωνο μιλητή. Ή παίρνουμε κάποιον που είναι πολύ καλό στη δουλειά του και μέσω μεταφραστή διερμηνία χάνουμε ένα 20% αλλά 70% βγαίνει προς τα έξω, υπάρχει επικοινωνία. Τι κάνουμε. Εκφράζω έτσι μεγαλόφωνα τις σκέψεις μου. Λοιπόν, φέτος έχουμε προωθούμε την έννοιά μας για την ΚΕΠΑ. Είναι το έτος αυτό. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων παρουσιάζουμε το πρόγραμμα αυτό ανάπτυξη και παρουσιάζουμε προ τα κράτη-μέλη αυτά τα θέματα. Και προσφέρουμε κάποιε λύσει. Δεν είναι καλό να παρουσιάζει μόνο προβλήματα χωρί λύσει. Εμεί είμαστε εδώ να υπηρετήσουμε. Δεν θέλουμε να ξεφορτωθούμε τα προβλήματά μα στα κράτη-μέλη. Πρέπει να δίνουμε και κάποιε λύσει που μπορούν να λειτουργήσουν και θέλουμε να εφαρμόσουμε, να ελοπίσουμε κάποιες από τις λύσεις που προτείνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάπως καλύτερα τα πράγματα. Τίνουμε να προσλαμβάνουμε άτομα ίσως πρέπει να ζητήσουμε από ευρωπαϊκές δυνάμεις να δώσουν στελέχη για τη Σομαλία. Πρέπει να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία στη στελέχωση. Οι άνθρωποι είναι το άπαν στις αποστολές. Ο φορέας είναι τόσο καλός όσο και τα στελέχη του. Λοιπόν, ακούστηκαν κάποια άλλα σχόλια. Ε, αυτό που παρουσιάσατε, ε, αναφερθήκατε στη Λιβύη. πώς εκτελεί την εντολή η αποστολή. Αυτά τα θέματα που θίξατε δεν καλύπτουν από την εντολή. Εμείς έχουμε σαν καθήκον να δούμε τι γίνεται με την ε, πολιτική ακτοφυλακή. Δεν είναι ευθύνη της αποστολής αυτό που αναφέρατε. Κοιτάξτε, ίσως κάνουμε μικρή διαφορά εκεί. Το πρόβλημα σε άλλα μέρη είναι να βρούμε τους σωστούς συνεργάτες. Δεν θέλουμε να εκπαιδεύσουμε κάποιους που είναι τόσο καλοί, να κάνουν λιγότερο καλό πράγματα, πιο αποτελεσματικά. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους ντόπιου, όπου θέλουμε σταθερά μέλη, συνεπή μέλη. Αν δείτε για την εντολή για τη Λιβύη και τι έκανε η αποστολή βάσει της εντολής, νομίζω ότι καλύψαμε τα περισσότερα στοιχεία της εντολής. Λοιπόν, εγώ λογοδοτώ και προσπαθώ να ενημερώσω 28 κράτη-μέλη που μου δώσαν την εντολή. Αυτό θα κάνετε φέτος, αυτό δεν θα κάνετε. Κάνετε αυτά και δεν θα κάνετε εκείνα, μου λέει η εντολή που μου δίνουν τα 28 κράτη-μέλη. Σημειώνω αυτά που είπατε όμως. Κατανοώ τα σχόλια που κάνατε για κάποιες αποστολές, όχι μόνο για τη Λιβύη, όπως και στο Μάλι, Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει η εντολή να κάνουμε. Ανάλογα με την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση ασφαλείας, σημειώνω τα σχόλιά σας και σε ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να έχουμε ειλικρινή ε, ανταλλαγή απόψεων. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Ε, οι Γυριγινή και οι κάτοικοι του Μάλι και οι Λίβγοι μου λένε «Κοιτάξτε, είναι λαμπρή η δουλειά που κάνετε και οι άνθρωποι σας υπέροχοι». Εντάξει, ίσω ο εγωισμό μου θέλει να τα πιστεύω αυτά. Αλλά ε, εδώ είναι η χρησιμότητα τη Επιτροπή σα. Καλό να ακούσω και τι επικρίσει. Είναι καλό να μιλάω και με τα κράτη-μέλη και με άλλου οργανισμού και έτσι ανακαλύπτω ποια είναι η αξία μα. Η εντολή μα ταιριάζει με την κατάσταση. Έχουμε σωστή εστίαση στι προσπαθίε μα. Ευχαριστώ ε, για τα ειλικρινή σα σχόλια. Και αυτά που είπατε, κυρία Πρόεδρε, στην ε, η Γεωργία Στη Γεωργία έπαιξε σημαντικό ρόλο η επικοινωνία. Η Γεωργία επικοινώνησε σωστά το ρόλο που, παρουσίασε το ρόλο που παίζουμε εκεί. Θα παραμείνει η αποστολή. Ένα προσωπικό σχόλιο, αν επιτρέπετε. Πρέπει η αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω τη Γεωργία να μην γίνει ένα κομμάτι του προβλήματο. Γιατί το λέω αυτό. να ε, εμποδίσουμε τα διάφορα εμπλεκόμενα κόμματα και μέρη να συμμετάσχουν στις διεργασίες επιλύσεως του προβλήματος. και να παρεμποδίζουμε την επίτευξη πιο μακροπρόθεσμης λύσης. Και να αποφεύγουν να βρουν μια συμφωνία μεταξύ τους τα εμπλεκόμενα μέρη. Λιβύη, Αφγανιστάν λοιπά. Πόσο επιτυχείς είμαστε, δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω ποια η κατάσταση θα ήταν εκεί αν δεν ήμασταν εμείς εκεί. Δύσκολο να το κρίνει κανείς αυτό. Αν δεν περάσει κάποια δεκαετία όπως και στις χώρες μας. Όταν μιλάμε στην όμευση κράτος δικαίου κλπ. Αυτά δεν συμβαίνουν μια ανοιχτή οι βελτιώσεις. Και έχουμε πολύ χαμηλή βάση. Έχουμε δύσκολη κατάσταση στην αρχή σε αυτές τις χώρες, η πολύ λίγη χρηματοδότηση. Είναι πολύ δυσχερείς οι καταστάσεις, πάρα πολύ περίπλοκες. Αν δεν ήταν οι αποστολές εκεί, τι θα γινόταν. Αν δεν ήταν εκεί, η αποστολή στη Γεωργία κάθε επαφή αφήνει ίχνος. ακόμα και αν μιλάμε με εκείνους που δεν δέχονται τις προτάσεις μας. Φυτεύεται, ίσως και έμεσα στο μυαλό τους και ίσως κάνει τη διαφορά. Αν δεν είμαστε εκεί, εάν δεν αναφέρουμε κάποια καλή πρακτική, δεν θα ακούσουν κάποιες καλές συμβουλές αυτοί οι άνθρωποι. Όσον αφορά τη Σομαλία, δίκιο έχετε. Οργανωμένο έγκλημα. Είναι οργανωμένο έγκλημα. Λαθρεμπόριο, πειρατεία, παράνομη αλληλεία, διάφορες παράνομες δραστηριότητε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζουμε ότι σε τοπικό επίπεδο μπορεί να αρχίσουν να, να αναπτύσσουν αντοχή και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ντόπιοι. Η Σομαλία θα ήταν στο επίπεδο του Αφγανιστάν εάν επέτρεπε η αποστολή μας να εκπαιδεύσουμε την τοπική αστυνομία. Πρέπει λοιπόν να γίνονται μετρημένες οι κρίσεις. Εάν έχει 50% στελέχωση η αποστολή τώρα, πρέπει να επεκταθεί η ε, ενταλή για να πετύχουμε το στόχο. Κινείται και ο ΙΕ σε αυτά τα πλαίσια. Δεν πρέπει να δημιουργούνται α, προσδοκίες για αυτοφυλακή κλπ. Και, και μετά να μην μπορούμε να τα αποκριθούμε. Πρέπει να υπάρχει σωστή στελέχωση στις αποστολές. Δεν αναγνωρίζουν οι εγκληματίε έντολε, όπω και το έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα. Αλλάζουν και τι τακτικέ του οι εγκληματίε πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι κάλυψα τι ερωτήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να υπερασπιστώ την Ευρωπαϊκή Εντολή, να σας πω ότι τα θέματα που αφορούν τη γεωργία είναι περίπλοκα. Και δεν νομίζω ότι θα βρισκόταν λύση εν απουσία της Ευρωπαϊκής Αποστολής. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ επίσης που δώσατε το χρόνο σας και ήρθατε. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, τις επιλοφορίες που μας δώσατε, όλα τα στοιχεία που δώσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δουλειά που κάνατε και εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάδελφοι, και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο, που είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο για τις διαστημικές δυνατότητες, για την ασφάλεια και την άμυνα. Και αυτό το σημείο, με μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω τον κύριο Φιλίπ Γρινέ, που είναι Διευθυντής Διαστημικής Πολιτικής του Κοπέρνικου και της Άμυνας τη Γενική Διεύθυνση Grow της Κομισιόν. Ο κ. Μουνέ είναι μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας Κομισιόν για το EDIDP, τον κανονισμό αυτό. Για πρώτη φορά το πρόγραμμα θα δώσει στην Ένωση τα απαραίτητα μέτρα για να υποστηρίξει την ανάπτυξη ε, χερσαίων, ε, θαλάσσιων και διαστημικών δυνατοτήτων για την ασφάλεια και την άμυνα η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει μεγαλύτερο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια και την άμυνα και πρότεινε να υπάρξει μια γενική διεύθυνση για αυτά τα θέματα στην Κομισιόν και άλλες δομές ε, και να συνεργαστεί με άλλες δομές ε, που αφορούν την άμυνα και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Σήμερα θα κοιτάξουμε τις δυνατότητες, ε, τις διαστημικές για την ασφάλεια και την άμυνα. Υπάρχει μια έκθεση που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2016 από τον κύριο Ζουντεύσκη. Ε, παρουσιαστήκε δύο χρόνια μετά ε, που διαπραγματευόμαστε τώρα το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα θέλαμε να κάνουμε, να παίξουμε το ρόλο μας, να δούμε που έχουμε φτάσει στην ασφάλεια και στην άμυνα και να ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Διευθυντής έχει το λόγο, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. κύριε Ευρωβουλευτές, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί το θέμα αυτό, γιατί η Κομισιόν πολύ πρόσφατα παρουσίασε το δημοσιονομικό πολιτέ πλαίσιο, όπου το διάστημα και η άμυνα ε, πήραν σημαντικά ποσά. Επιπλέον, από τις αρχές του Ιουνίου θα παρουσιάσουμε το κείμενο για την εφαρμογή της νέας στρατηγικής για το διάστημα. Λοιπόν, το θέμα το σημερινό αφορά τη δυνατότητα οι διαστημικές υποδομές να υποστηρίξουν την ασφάλεια και την άμυνα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορεί να απαντηθεί και με απλό τρόπο. Από αυτή τη στιγμή που το διάστημα χρησιμοποιήθηκε για την πλοήγηση ή για την ε, παρατήρηση της γης, αυτές οι δυνατότητες που είναι πολιτικής φύσεως στην Ευρώπη, ενώ σε πολλές άλλες χώρες είναι στρατιωτικής φύσεως, μπορούν να δώσουν πληροφορίες να δώσουν δεδομένα που έχουν ένα δυναμικό διτής χρήσης πολύ σημαντικό. Στο Κοινοβούλιο και στα κρατη υπάρχει μια τάση πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή υπέρ της διατήρησης της πολιτικής διαχείρισης του, των προγραμμάτων Κοπέρνικους και Γαλιλαίου. Πολιτικής διακυβέρνησης καλύτερα. Επίσης, αναγνωρίζουμε το σύνολο των δεδομένων ή των σημάτων που στα πλαίσια του Γαλιλαίου παίρνουμε. Έχουμε ειδικά κομμάτια για την ασφάλεια και για την άμυνα. Ενώ στον Κοπέρνικο χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο διάφορους αισθητήρε, ραντάρ, οπτικούς αισθητήρε, ε, υπέρυθρον επίσης, υπέρυθρους αισθητήρε, για να δούμε και στο μέλλον μάλλον θα έχουμε και μη διαστημικούς αισθητήρε, όπως ε, οι πλατφόρμες υψηλού, σε υψηλό, μεγάλο ύψος. Όλοι αυτοί οι αισθητήρε δίνουν εικόνες, δίνουν γεωγραφικές θέσεις και συνεχεία αυτά τα δεδομένα μπορούν να μας βοηθήσουν και για την ε, πολιτική ασφάλεια, αλλά και για την ε, στρατιωτική ασφάλεια και για την άμυνα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι κάποιες υπηρεσίες του Κοπέρνικου προς το παρόν ε, συνεργάζονται σε μεγάλο βαθμό με υπηρεσίες όπως ε, η Frontex ή όπως η υπηρεσία για την ασφάλεια στη θάλασσα, την ΕΜΣΑ. Στο μέλλον θα αναπτύξουμε μέσω εταιρικών σχέσεων με τη βιομηχανία μία προσέγγιση που θα μας επιτρέψει να έχουμε δεδομένα μεγαλύτερης ευκρίνειας που επικυροποιούνται πολύ πιο συχνά, δεδομένα υψηλής ακρίβειας, ε, που αν τα συνδυάσουμε τα δεδομένα από τα ραντάρ που έχουμε και με τα δεδομένα από το Κοπέρνικους ε, βέλειας 10 μέτρων, μπορούμε να φτάσουμε χάρη σε εταιρικέ σχέσεις με τη βιομηχανία με 30, ως τα 30 εκατοστά. Μπορούμε επίσης να δράσουμε μέσα σε μία ώρα, δηλαδή από τη στιγμή θα λάβουμε το δεδομένο. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να δούμε τι γίνεται με, την, με τις μεταστατικές ροές, με το λαθρεμπόριο κτλ. Αυτά τα δεδομένα δεν θα τα αποκτήσουμε για συγκεκριμένο σκοπό. Η χρήση που μπορεί να τους γίνει από τους τελικούς χρήστες εξαρτάται βεβαίως από το ενδιαφέρον τους και θα, τις, και θα τροποποιηθούν εν πάση περιπτώσει αυτές τις πληροφορίες ανάλογα με το ποιος τις χρησιμοποιεί. Οι στρατιωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ας πούμε ρύθμισης ας πούμε, που καταπολεμούν την παράνομη ασφάλ, ε, κτλ. Ε, η Επιτροπή σας ασχολήθηκε με την ε, διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην ασφάλεια και στην κυβερνοάμυνα. Δύσκολη διαφορά. Ε, είμαι υπεύθυνο για, για τα θέματα αυτά και κάναμε συζητήσει με τον αρμόδιο του Κοινοβουλίου. Και μερικέ φορέ η οριοθέτηση ανάμεσα στα δύο είναι δύσκολη και μπορούμε να περάσουμε εύκολα από το, να γλιστρήσουμε από το ένα στο άλλο. Σε ό,τι αφορά την παρατήρηση τη γη, επίση, όταν έχετε σε κάποια σύνορα για τη Frontex, ας πούμε, μια παρακολούθηση 30 με 50 εκατοστά με δυνατότητα επικαιροποίησης μέσα στην ώρα, σε περίπτωση ε, απειλής, ε, επίθεσης ε, στην ε, ασφάλεια της Ευρώπης, αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμα. Ποια είναι τα μεγάλα προγράμματα, τα μεγάλα συστήματα σήμερα, που είτε έχουν τη δυνατότητα, είτε παράγουν δυνατότητες γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε υπηρεσίες από την βιομηχανία. Ποια είναι τα μεγάλα λοιπόν συστήματα που θεωρώ ότι έχουν μεγάλη σημασία για την άμυνά μα. Καταρχάς όλοι ξέρουν το Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίος με 22 δορυφόρους και δύο ακόμα που θα είναι σε λίγο λειτουργική αποτελεί ένα σύστημα πλοήγησης το οποίο είναι πολύ πιο καλό από την τρέχουσα χρήστη του αμερικανικού, τρέχουσα εκδοχή του αμερικανικού GPS. Το, ο Γαλιλαίο από την αρχή είχε ένα σύστημα IPRS δημόσιο που είναι διαθέσιμο για τους εγκεκριμένου χρήστες, δηλαδή τις εθνικές αρχές γενικά, που είναι πάρα πολύ αξιόπιστος σε ό,τι αφορά την, το σήμα και το σήμα είναι πολύ ακριβές. Είναι σαφές ότι και αστυνομικέ αρχές, αλλά και οποιοδήποτε οποιαδήποτε αμυντικός φορέας θα μπορούσε, και αυτοί είναι οι βασικοί μας πελάτες εξάλλου, να χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα PRS. Για τον Κοπέρνικο έχουμε πριν από 15 μέρες ξεκινή, ε, δρομολογεί στον 7ο δορυφόρο. Η διαφορά μεταξύ του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου είναι ότι στους 22 και ως ονούπο 24 δορυφόρους του Γαλιλαίου όλοι οι δορυφόροι μοιάζουν με τον πρώτο. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε ε, σήματα από όλο τον πλανήτη, ούτω ώστε να ξέρουμε με αρκετά μεγάλη ακρίβεια τι γίνεται. Στο Κοπέρνικο, ο κάθε από τους 7 ε, δορυφόρους ανήκει σε διαφορετική οικογένεια, σε διαφορετική κατηγορία. Ε, εξού και η διαφορά σε σχέση με το αμερικανικό σύστημα. Γιατί ε, σε διαφορετικές πλατφόρμε έχουμε διαφορετικούς αισθητήρε. Ε, και να σα τονίσω κάτι που μάθαμε εμεί όταν α, ξεκινήσαμε τον Κοπέρνικο. Μπορούμε να διασταυρώνουμε δεδομένα. Δηλαδή, όταν έχουμε όχι μόνο οπτικά δεδομένα, αλλά και υπέρ, υπέρ υπέρυθρα, η υψομέτρου ε, έχουμε διαφορετικές πληροφορίες και αν διασταυρώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες φτάνουμε στο να έχουμε προϊόντα τα οποία είναι καλύτερα από την, την απλή ε, συσσόρευση ε, μεμονωμένων δεδομένων. Το Κοπέρνικους έχει και μία διάσταση για την ασφάλεια και συνεργάζομαστε εδώ πέρα ε, με, το, με τη Frontex και την Emsa και με το ΣΑΤΣΕΝ και στα πλαίσια του ΣΑΤΣΕΝ ε, παίρνουμε πληροφορίες για τις δράσεις που γίνονται στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ως υπάρχει η δυνατότητα τώρα να αυξήσουμε τις, τη διάσταση αυτή της ασφάλειας Παραθετικά να σας πω ότι τα μεγάλα χαρακτηριστικά του Κοπέρνικου είναι ότι προωθεί μέσω ελεύθερων δεδομένων, ε, δωρεάν δεδομένων, την ε, δημιουργία ενός οικοσυστήματος, ούτως ώστε διάφορες ε, εφαρμογές και διάφορες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά αυτή την πρώτη λοιπόν τα δεδομένα και να υποφελούνται ας πούμε. Αυτή η ανοιχτή πολιτική δεδομένων, τα ελεύθερα δεδομένα, δεν ισχύει στην περίπτωση του συστήματο που ασχολείται με την ασφάλεια. Όπου καταλαβαίνω ότι κάποια προϊόντα τα οποία προκύπτουν από αυτά τα δεδομένα φυσικά έχουν πολύ ευαίσθητο χαρακτήρα και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο καθένα. Στην πρόταση κανονισμού το που εκπονούμε αυτή τη στιγμή, κάποιε ιδέε ακούστηκαν, δεν μπορώ να σα πω τώρα εάν το σώμα των επιτρόπων θα τι κρατήσει ή όχι, αλλά υπάρχει η δυνατότητα, η δυνατοτητα να δημιουργήσουμε εταιρικέ σχέσει με τη βιομηχανία, ούτω ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα δεδομένα των δορυφών του Κοπέρνικου με τα δεδομένα άλλων πηγών και να φτιάξουμε μεγαδεδομένα, με, με μεγαλοδεδομένα της βιομηχανίας ή ε, να συνδυάσουμε και τις δορυφορικές ικανότητες των κρατών μελών και με αυτό το νέο τύπο αισθητήρων που ονομάζουμε hubs, ε, ε, που είναι συστήματα, πλατφόρμες υψηλού ε, υψομέτρου, που είναι σαν αερόστατα και μπορούν να μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από μια περιοχή και που θα οδηγήσουν σε επανάσταση. Γιατί, λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό υψόμετρο, παρότι το ονομάζουμε υψηλού υψομέτρου, σε σχέση με τους δορυφόρους που είναι ακόμα πιο ψηλά, μπορούμε να δούμε δεδομένα σε βίντεο. Δεν θα είναι τεροχρονισμένα αυτά τα δεδομένα, θα είναι δηλαδή πραγματικού χρόνου. Επομένως, το σύνολο αυτών των συστημάτων θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνεκτικό όλο. Και χάρη στην, στο συνδυασμό αυτών των δεδομένων έχουμε ένα καλό τελικό προϊόν, που είναι πολύ ανώτερο από αυτό που θα είχαμε ε, αν είχαμε μεμονωμένα αυτά τα συστήματα και δεν τα είχαμε όλα. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα Space Surveillance and Tracking, SST. Ξέρετε πολύ καλά ότι πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες ο, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πέντς ζήτησε να ξανασκεφτούν οι Αμερικανοί να υπάρχει ρύθμιση του, της κυκλοφορίας των δορυφόρων. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εκεί. Αυτό ε, θα δημιουργήσει τεράστιες δυσκολίες, γιατί για να ρυθμίσουμε την, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο τους δορυφόρους θα πρέπει ε, οι ρυθμιστικές αρχές να είναι παγκόσμιες. Ε, αλλιώς δεν λειτουργεί. Γιατί αναφέρω αυτό το πρόγραμμα SST. Γιατί η πιο βεβαρημένη αποκίνηση τροχιά, σε αυτήν θα πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται με τους δορυφόρους και να μην ε, συγκρουστούν ας πούμε οι δορυφόροι ε, με διάφορα θράψματα. Ε, μιλάμε για ύψος 800 με 900 χιλιόμετρα περίπου. Αν κοιτάξετε ποιο είναι το υψόμετρο των βαλιστικών πυράβλων που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες χώρες που έχουν τέτοιους πυράβλους, βλέπουμε ότι αυτοί οι πυραβλοί γενικά κινούνται μεταξύ 500 μέτρων και 2 χιλιόμετρων. Ε, κανονικά μιλάμε για ένα σύστημα τηλεσκοπίων και ραντάρ, ούτως ώστε οι δορυφόροι μας, οι υποδομές μας να μπορέσουν να συνεχίσουν να ε, υπάρχουν χωρίς να υποστούν ζημιές από τα θράψματα. Θα, για να έχουμε λοιπόν αυτά τα πετούμενα που δεν θα είναι ούτε δορυφόροι ούτε θράψματα, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προσπάθειες. Επομένως υπάρχει ένα νέο πεδίο συνεργασίας εδώ με τα κράτη-μέλη, δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θα πρέπει να προστατεύσουμε τις υποδομές μας, αλλά θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο εναέριο σύστημα άμυνας των κρατών μελών. Και όταν, λέω, όταν μιλάω για αυτό το σύστημα εναέριας ε, Μιλάμε για το, και για τις μεγάλες συμμαχίες, όπως το ΝΑΤΟ. Γιατί ξέρετε ότι το ΑΓΟΑΞ που ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες και ορισμένοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να βρεθεί η διάδοχη κατάσταση με άλλου τύπου ραντάρ που δεν είναι σε σκάφη. Εδώ μπορούμε να δούμε μια συνέργεια ανάμεσα στα δορυφορικά προγράμματα που σκοπό έχουν να τελειοποιήσουν τα συστήματα δορυφορικής προστασίας με το κατόπιν, ας πούμε, αιτήματος ενός κράτους μέλους, ε, με μια διάσταση βαλιστική, ας πούμε. Συνδυασμένη με βαλιστική διάσταση. Και κάτι που είναι το γενάστε είναι το πρόγραμμα Golfstat.com θα ξεκινήσει πώς. Θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δομές, όλες τις δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη μαζί, σε ό,τι αφορά τους δορυφόρους τηλεπικοινωνιών και θα προσθέσουμε αυτά που θα μας προτείνει η βιομηχανία. Φυσικά τα κράτη-μέλη δεν ενδιαφέρονται όλα το ίδιο για αυτό το πρόγραμμα. Παραδοσιακά, τα κράτη-μέλη που έχουν ε, μεγαλύτερη στρατιωτική δραστηριότητα. Ε, τα μεγάλα κράτη-μέλη που έδρασαν στο εξωτερικό της Ευρώπης φυσικά έχουν αυτές τις δυνατότητες. Αυτά είναι 5, 6, 7 και είμαστε 28 στην Ένωση. Επομένως αυτό το πρόγραμμα θα επιτρέψει στο να χρησιμοποιήσουμε ή μάλλον όλοι μαζί τι δυνατότητέ μα και να δώσουμε δυνατότητε σε κρατη που δεν διαθέτουν. Ακόμα και τα κρατη που έχουν αυτέ τι δυνατότητε, μιλάμε για γεωστατικού ε, δορυφόρου. Έχετε αυτό το ε, δορυφόρο σα κάπου, α πούμε, στην Ευρώπη ή στην Αφρική. Αν έχετε όμω ένα θέατρο δράση, το οποίο βρίσκεται στην ε, Κορέας, στην κερσόνησο της Κορέας. Ή αν θέλετε, κάποια δράση ας πούμε, στον ειρηνικό, δεν μπορείτε να μετακινήσετε τον δορυφόρο σας. Εκεί εξαρτάστε από τις, τα συμβόλαια με τη βιομηχανία ή με τους συμμάχους εντό εισαγωγικών που μπορεί, ναι, μπορεί να μην σας δώσουν πρόσβαση στον δορυφόρο σας εκεί που θέλετε, στο σημείο που θέλετε. Και που αν σας δώσουν φυσικά πρόσβαση στον δορυφόρο τους, φυσικά θα, έχετε πρόσβαση και στις πληροφορίες που περνούν από αυτό το ε, δορυφόρο. Το τρίτο σημείο, πολύ σημαντικό, εδώ είναι ότι στα πλαίσια αυτών αμυντικών προγραμμάτων μιλάμε όλο και περισσότερο για τα οχήματα, ειδικά για αναγνωριστικά drones. Τα drones, εκτός του ότι πρέπει να, είναι, να είμαστε θέση να τα κατασκευάσουμε και προς το παρόν, πέρα από τους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς δεν έχουμε φτάσει στο ίδιο, σε, σε αυτό το τεχνολογικό επίπεδο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε γρήγορα. Τα drones εξαρτούνται από δύο πράγματα. Καταρχάς, από σήματα ασφα... ε, από σήματα κυβερνοασφάλειας πολύ σημαντικά. Ούτω ώστε να μην πάρει κάποιο τον έλεγχο ας πούμε, το, του drone σας ή να μην του δώσει λάθος πληροφορίες. Και δεύτερον, από τις, ε, τηλεπικοινων... τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους. Συχνά μιλάμε για drones που χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι και που τα πιλωτάρουν από μια βάση στη Μασαχουσέτη, ας πούμε. Ε, όταν χρησιμοποιούνται στο Αφγανιστάν ή στην Αραβική Χερσόνησο, φυσικά τα σήματα θα πρέπει να φύγουν από τη Μασαχουσέτη για να φτάσουν εκεί που βρίσκονται και που θα χρησιμοποιηθούν οι drones. Και μιλάμε για σήματα ε, Και όταν το drone είναι αναγνώριση, ε, βλέπει κάτι και εσείς του ξαναστέλνετε πίσω το, το σήμα. Μιλάμε για τεράστιες αποστάσεις. Ε, λίγα είναι τα κράτη μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείες που έχουν παγκόσμια κάλυψη. Επομένως, ε, μια άλλη από τις πρωτοβουλίες αυτού του προγράμματος είναι να μην αντικαταστήσουμε αυτό που υπάρχει ήδη, αλλά να προσφέρουμε αυτό που δεν υπάρχει, ε, τον ε, κρίκο της που λείπει, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση να έχει με ασφαλείς ε, επικοινωνίες με όλους, αλλά και στα δεύτερα, στα, στο επίπεδο της ΚΠΑ, όποιος και είναι ο λόγος της δράσης και ο στόχος της δράσης, όπου και αν λαμβάνει χώρα αυτή η δράση, να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις δυνατότητε των κρατών μελών ή αν δεν υπάρχουν αυτές, στις ευρωπαϊκές δυνατότητε. Τελευταίο σημείο. Ξέρετε και σας το είπατε κυρία Πρόεδρε, ότι αυτή τη στιγμή είναι υποσυζήτηση το project IDEP, που στο μέλλον θα οριστικοποιηθεί ε, το... με σκοπό, ας πούμε, α, το, το, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που θα έχει ένα επιρσιακό κομμάτι και ένα κομμάτι για την άμυνα. Μέχρι στιγμής υπάρχει μια προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα. Το άλλο κόμμα σχέδιο ήταν η έρευνα μάλλον. Επίσης, πολύ σημαντικό, στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα έχουμε ένα παράδειγμα, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να καταδείξουμε ότι υπάρχει ανάγκη για δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προωθήσει συνεργατικά project. Ε, ονομάζεται Οκεανή 2020, ε, όπου συμμετέχουν 10-15 κράτη-μέλη και πολλές εταιρείες και που σε σκοπό έχει, όπως βλέπετε και από το όνομά του, να μας δώσει δυνατότητες ε, θαλάσσιας εποπτείας για λόγους ασφάλειας ή άμυνας. Αυτό το project είναι ερευνητικό ακόμα. Αυτό το πρόγραμμα είναι ερευνητικό και θα στηριχθεί στους πόρους των κρατών μελών, ειδικά της Ιταλίας, ε, του κόσμου, Skymer, ε, εικόνες ε, μέσω ραντάρ ή τους δορυφόρους του Κοπέρνικους. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια συμπληρωματικότητα σε αυτά τα project. Καταρχά και δημοσιονομικά. Δεν έχει νόημα απλώ με δύο φορέ ερευνητικά προγράμματα όταν τρέχει ήδη ένα. Θα πρέπει ίσω να τροποποιήσουμε τι ανάγκε του ερευνητικού προγράμματο. Αλλά δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε πάντα από, πάλι από το μηδέν. Όταν έφτασα εδώ σε αυτή τη δουλειά, μου είπαν ότι υπήρχαν ήδη συστήματα παρατήρηση τη γη σε επίπεδο κρατών μελών. Υπήρχε και στις, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιαπωνέζοι είχαν και αυτή το δικό τους. Το ερώτημά μου ήταν λοιπόν γιατί να φτιάξουμε και εμείς επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για έναν απλό λόγο. Γιατί δεν υπάρχει κανένα τέλειο σύστημα. Παρά ότι το Κοπέρνικο είναι το καλύτερο από όλα. Γιατί ποτέ δεν είσαστε σίγουρος ότι, ο δορυφόρος σας μαζί με τον σωστό ε, αισθητήρα ε, την κατάλληλη στιγμή βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο. Όσο περισσότερα συστήματα παρατήρησης έχετε, Όσο περισσότερους αισθητήρε έχετε που είναι συμβατοί και με τους οποίους, στους έχετε πρόσβαση, έχετε μεγαλύτερη σιγουριά τη στιγμή που γίνεται κάτι. Το, ή το δικό σας σύστημα, ή το σύστημα των συμμάχων σας, ή το σύστημα ενός κράτους μέλους στην περίπτωση της Ευρώπης, θα είναι στο κατάλληλο σημείο το σημείο που μας ενδιαφέρει. Αυτή λοιπόν η συνέργεια των συστημάτων πρέπει να ξεκινήσει από τη στιγμή της, του σχεδιασμού και της έρευνας. Ακριβώς γι' αυτό νομίζω ότι θέλουμε να υπάρχει και συνέχεια και εξέλιξη των ευρωπαϊκών συστημάτων. Να δούμε επίσης πώς θα εξελιχθούν οι ανάγκες μας και να διασφαλίσουμε και την αυτονομία μας. Αυτή είναι η πρόκληση. Όπως το είπα και στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων. Αν έχετε ανάγκη ένα τέτοιο δορυφόρο από μια εταιρεία τη στιγμή χ που ανήκει στο κράτος γ, δεν σημαίνει ότι έχετε πάντα την πρόσβαση που θέλετε στον ε, δορυφόρο. Ακόμη και εντός της Ευρώπης. Στο gov.satcom θα πρέπει να λύσουμε το θέμα της ιεράρχησης των ετοιμάτων που θα τίθενται. Και για τα θέματα αυτά, DG Grow θα πρέπει να συμβουλευθώ τους συναδέλφους της υπηρεσίας εσωτερικής δράσης που αυτοί θα αποφασίσουν γιατί αυτοί διαχειρίζονται τα προγράμματα. Εγώ τους δίνω τα εργαλεία και το εγχειρίδιο με τις οδηγίες αλλά αυτοί θα το χειριστούν. Το τελευταίο σημείο έχει πει για την, ε, έχουμε πει για την ε, συνέχεια και την αυτονομία για θέματα ασφάλειας. Υπάρχει μια υποχρεωτική συνεργασία μεταξύ των ε, αναγκών μας στρατιωτικής ασφάλειας και πολιτικής ασφάλειας. Οι ψηφιακοί δορυφόροι παράγουν τα μηδενικά και τις μονάδες. Μετά οι επεξεργαστές μας θα μας δώσουν τις προφορίες. Είτε είμαι στρατιωτικός με έναν τρόπο, είτε είμαι πολιτικό προσωπικό με άλλο τρόπο. Αλλά το σύστημα από την αρχή θα πρέπει να ε, ε, μου δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσω και τα δύο συστήματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και υπογραμμίζω ότι βασιζόμεθα πολύ στα πλαίσια των διαδικασιών του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου στην λήψη υπόψη από πλευρά του Κοινοβουλίου αυτών των δύο κριτηρίων. Ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια στι προσπάθειέ μα, αλλά και ότι πρέπει να είμαστε αυτόνομοι στη δράση μα. Γιατί η πρόσφατη πείρα κατέδειξε σε έναν άλλο τομέα. Να τον αναφέρω. Αν και αφορά κυρίως την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε συνεργασίες που αποφασίζονται ή αμφισβητούνται από τρίτες χώρες. Όπως ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα ο Λευκός Οίκος ακύρωσε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της γης για την κλιματική αλλαγή. Και ένα τμήμα του Κοπέρνικου για την κλιματική αλλαγή δεν είχε αναπτυχθεί γιατί θέλαμε να αξιοποιήσουμε το αμερικανικό σύστημα που ήδη υπήρχε. Και τώρα δεν υπάρχει και θα πρέπει να αναπτύξουμε το δικό μας. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα με τα υπάρχοντα συστήματα. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Και δεν μπορούμε να βασιζόμεθα σε συστήματα που δεν εξαρτώνται από εμάς. Πρέπει να διασφαλίσουμε κάποια στιγμή την αυτονομία μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Και τώρα το λόγο έχουν οι συνάδελφοι. Ο Μάικλ Γκάλερ θα είναι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ για αυτή την επισκόπηση. Για την κατάσταση αυτή τη στιγμή και τους στόχους μας. Όλοι παρακολουθούμε αυτές τις δραστηριότητες όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το διάστημα. Είναι θέματα όπου εργάζεται ιδιαίτερα και ο συνάδελφος Στογεύσκη, εδώ πίσω μου. Είπατε τώρα ότι οι Αμερικανοί δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Άρα πρέπει πολλά να τα προωθήσουμε εμείς και να βασιστούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Και επειδή έτσι είχε η κατάσταση και επειδή παρόλα αυτά έχουμε επαρκείς πόρους με βάση το πρόγραμμα όπως ανακοινώθηκε πρέπει να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας και ελπίζω να το καταφέρουμε φροντίζοντας ωστόσο να μην υπάρξουν επικαλύψεις. Σε τομείς που ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό και τα αναφέρατε κι εσείς. Ξέρω. Στο ότι σε κάποιους τομείς υπάρχουν και καταστάσεις ανταγωνισμού. Τριβές. Ποιος πρέπει να κάνει τι. Αν θα πρέπει να γίνει κάτι με τον α ή τον β τρόπο. Αλλά δεν πρέπει να εμποδίσουν όλα αυτά την βελτιστοποίηση της συνεργασίας. Επειδή έχουμε πολλά καθήκοντα, τονίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσω του ESA. Δεν πρέπει να τα επικαλύψουμε, να κάνουμε κάτι παράλληλο. Να επικεντρωθούμε σε αυτά που ακόμη δεν τα έχουμε. Τα κενά που πρέπει να καλύψουμε. Και να προωθήσουμε τη συνεργασία με οργανισμούς που δεν έχουν τα ίδια καθήκοντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή χρήση των πόρων. Με τον βέλτιστο τρόπο. Και ελπίζω λοιπόν να συνεργαστούν σωστά όλοι οι εμπλεκόμενοι και από πλευράς μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να καθορίσουμε τις ευθύνες και τα καθήκοντα του καθενός. Σας διαβεβαιώ ότι ούτως ή άλλως θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι ακόμη για την DG Defense και τον ε, αεροναυτικό τομέα, τον αεροναυπηγικό τομέα. Άμυνα και διάστημα. Τι γίνεται γι' αυτά. Γιατί ε, τα στηρίζω ιδιαίτερως και ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάικλ. Ο κ. Τρογεύσκη έχει το λόγο. Λοιπόν, θα αναφερθώ στο σημείο που αναφέρθηκε στην αρχή της συζήτησης. Η συζήτηση έχει λάβει χώρα και αφορά τους δορυφόρους. Και είχαμε συζητήσει για πρώτη φορά τους δορυφόρους τότε στην Επιτροπή μας. Έχουμε τέσσερα στοιχεία για αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ζητήσουμε την κατασκευή, να την ύπαρξη κάποιων οικονομικών εγγυήσεων μακροπροθέσμων. Υπογραμμίσαμε λοιπόν ότι η δραστηριότητα δεν ήταν αρκετή στον τομέα αυτό. Δεν υπήρχε καλή συνεργασία και εν ώψη της συγκεκριμένης τεχνολογίας έπρεπε να αναφερθούμε στις δημοσιονομικές προοπτικές. Είχαμε συμφωνήσει επί του επιδιωκόμενου στόχου τότε. Σήμερα πρέπει να πω ότι υλοποιούμε το στόχο 1. Θα υπάρχουν οικονομικές εγγυήσεις μέχρι το 2027 ο προπολογισμό θα, θα αυξηθεί από 12 σε 16 δισεκατομμύρια και θα εξασφαλίσουμε και τη βελτίωση ε, της καταστάσεως της έδρας στην Πράγα, όπου υπήρξαν κάποια οικονομικά προβλήματα και προβλήματα προσλήψους ε, προσωπικού. Τέλος, ο δεύτερος στόχος είναι η τεχνολογική πρόοδος. Ξεκινήσαμε μέσω των πληροφοριών και εξαρτώμεθα λοιπόν για, εξαρτώμεθα για την εκτόξη των δορυφόρων από ρωσικούς πυράβλους. Θα έπρεπε να έχουμε δικούς μας ε, ε πυράβλους και κάποια φορά είχαμε κάνει και λάθος εκτόξευση, είχαμε βάσει σε λάθος τροχέα δορυφόρους. Είχαμε αποτελέσματα τώρα πολύ ικανοποιητικά. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι τώρα Έχουμε τους δύο στόχους όσον αφορά την παρατήρηση των θαλασσών ε, και είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι. Έχουμε και τον πύραυλο Vega, τον Αριάν, τον Αριάν 5, που λειτουργούν αυτοί οι πύραυλοι και θα φτάσουμε και στην κατασκευή του Αριάν ε, 6. Είναι ο μεγαλύτερος πύραυλος και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 2020. Μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη στο συγκεκριμένο πλαίσιο θα είναι πολύ πιο αυτόνομη, πολύ πιο ανεξάρτητη από ό,τι μέχρι πριν από τρία χρόνια. Χαίρομαι μπορώ να πω ότι στα πλαίσια του δικού μας ευρωπαϊκού συστήματος πλοήγησης έχουμε ήδη 20 δορυφόρους σε τροχιά. Να υπενθυμίσω ότι έπρεπε να έχουμε 30 δορυφόρους. Στα πλαίσια των 30 πρέπει να έχουμε και 5-6 σε απόθεμα θέλετε. Είμαστε πολύ κοντά προς το τέλος του προγράμματος και είμαστε πεπισμένοι ότι μέσω υποστήριξης ε, έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στην ολοκλήρωση των προσπαθειών. Τώρα το τρίτο στοιχείο που απαιτείται για το πλαίσιο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ε, διαφημιστικές δραστηριότητες, προωθητικές δραστηριότητες. Υπάρχουν δαπάνες ε, από Κοπέρνικος σε Γαλιλαίο, και οι δαπάνες θα πρέπει να, χρησιμοποιούνται και στην ενημέρωση. Θα πρέπει οι καταναλωτές και οι πολίτες να ξέρουν ε, επίσης και τι προγράμματα μπορούμε να τους προσφέρουμε μέσω των δορυφόρων και να χρησιμοποιούνται υπηρεσίες. Αυτό τελευταία έγινε πολύ καλά, η ενημέρωση για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Σας συγχαίρω λοιπόν κύριε Διευθυντά είναι ορατή η προσπάθεια διαφήμισης και ενημέρωσης, είναι ορατή, απτή ε, η πρόοδος που έχει σημειωθεί. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τέταρτο ε, στοιχείο που δεν λειτουργεί ακόμα και είναι πρόκληση για μας. Καλύτερη διασύνδεση με την ιδιωτική αγορά στα πλαίσια της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα που αναφέρατε. Θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια των δαπανών και των υπηρεσιών να έχουμε μια συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων. Και εδώ έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, αλλά πάντα είναι μέτρια η πρόοδος και δεν μας ικανοποιεί. Τέλος, κάτι που συνδέεται με το μέλλον, είναι τα απόβλητα και τα θαύματα ε, στο, διάστημα. Υπάρχουν ε, δεκάδες χιλιάδες αρκετά μεγάλα αντικείμενα που ε, μολύνουν, αν θέλετε, ρηπαίνουν τις τροχές που πάνε οι δορυφόροι. Και επίσης είναι και απόβλητα που είναι από τεχνολογικά αντικείμενα που χρησιμοποιούμε πλέον. Πρέπει να κάνουμε κάποιες προσπάθειες να... Κάναμε προσπάθειες να τακτοποιήσουμε κάπως την κατάσταση, αλλά με πολύ μικρή επιτυχία. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ε, φορέων, με τη ΣΥΠΑ, με την Κίνα, με τους Ιαπωνέζους. Πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία με αυτές τις τιμικές δυνάμεις. Οι Κινέζοι προσπάθησαν προσπάθησαν έκανα κάποιες προσπάθειες αλλά με τις προσπάθειες που έκαναν να καθαρίσουν το διάστημα έβλαψαν κάποιους δορυφόρους που ήταν λειτουργικοί Χρειάζεται λοιπόν ένα διαστημικό νοικοκυριό, αν θέλετε, να βάλουμε μια τάξη στο διάστημα. Και τέλο είναι τα μη επανδρομένα επτάμενα χήματα τα drone. Υπάρχουν drones που κοστίζουν 70 ευρώ, πολύ φθηνά, ε, και υπάρχουν και άλλα που μπορεί να γνωρίζουν να κοστίζουν 70 ε, εκατομμύρια ευρώ και μας επιτρέπουν να κινηθούμε σε ένα χώρο πολύ μεγάλου ύψους. Ο έλεγχος των drones που μπορούν να μεταφέρουν όπλα είναι ένα θέμα, που μπορούν να μεταφέρουν χημικά προϊόντα επί των αρρωσίμων γεών, αλλά να απειλήσουν και την Ευρώπη ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικότατο. Να σας υπενθυμίσω ότι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νομοθεσίες εθνικές που είναι ανεξάρτητες και δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ εθνικών νόμων τάξεων θα ήταν καλό να υπάρξει ένα συντονισμό για να μπορούμε να ελέγξουμε τα μη επανδρομένα αυτά σκάφη, τα drones, κάθε είδου και κάθε μεγέθου. Όσον αφορά τα τέσσερα βασικά σημεία που παρουσιάσαμε σαν προκλήσει και στόχου, οι τέσσερι στόχοι έχουν προχωρήσει λίγο πολύ. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις ε, προσπάθειες που κατεβλήθησαν και μπορούμε σε αυτή τη φάση να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το έργο των δύο υπηρεσιών και των άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με αυτούς τους δύο βασικούς ε, φορείς. Ευχαριστώ κύριε Στρογεύσκη. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος άλλος το λόγο, εκτός από την υποφανούμενη για μια ακόμη φορά. Καταρχάς, να πω, που απηχεί και την άποψη άλλων, και αφορά τα έξοχα επιτεύγματα μέχρι τώρα με το Κοπέρνικος και το Γαλιλαίος, με τα δύο συστήματα αυτά, σε όλες τις πτυχές, σε όλους τους τομείς, όχι μόνο τον αμυντικό, αναφερθήκατε σε συνεργασίες και τι μπορεί να επιτευχθεί με αυτές. Αυτό πολύ σωστά το παρουσιάσατε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα για την επικοινωνία επίσης. Ε, συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν και συνδέεται αυτό. Όπως τα προβλέψατε, ως Βρετανίδα Ευρωβουλευτής, θέλω να αναφερθώ και στα ατυχή γεγονότα, στο ατυχές γεγονός του Brexit. Εγώ ήμουν αντίθετη από την αρχή με το Brexit. Είναι μια θεματικά κακή ιδέα κατά την απόψή μου, αλλά εφόσον για την ώρα προχωράει και πρέπει να ζήσουμε με τις συνέπειες αυτού του γεγονότος, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημιές που δημιουργούνται από το Brexit. Δηλαδή, πιο πρόσφατα με το JCPRA είδαμε τη συνεχή ευθυγράμμιση του έργου αυτού υπό την ηγεσία Γερμανίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται, ότι είναι ένας τομέας όπου πολλά διακυβεύονται και θα θέλαμε και εγώ θα υποστηρίζα να υπάρξει στενή σχέσεις όπου να έχουμε αμοιβαία ωφέλη από τη σχέση. Κυρίως στο καυτό θέμα του PRS και του Γαλιλαίος. Σε όλα τα συστήματα και στο χώρο της, του διαστήματος κυρίως. Madam, um, as regards the uh, perspective... Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη προοπτική που αναφέρατε και την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν γίνει αυτή αποδεκτή, που θα επεκταθεί και μέχρι το 2027 η προσπάθεια, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε και πιο μακριά. Με το Κοπέρνικος, μαζί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, έχουμε συντάξει ένα έγγραφο. Μακροπρόθεσμο σενάριο είναι ο τίτλος του. Λόγω της διάρκειας ζωής των διαφόρων δορυφόρων και πρέπει να εξασφαλίσουμε και συνέχεια, όπως ξέρετε, πρέπει να σκεφτόμαστε και τι γίνεται πριν ε, από, πριν το τέλος του επομένου δημοσιονομικού ε, πλαισίου βέβαια ε, υπό την αίρεση της έγκρισης των αρχών του προπολογισμού. Ε, εκτιμώ αυτό που είπατε και πολύ. Δημιουργούμε ένα οικοσύστημα που βασίζεται σε συνεχή ροή δεδομένων. Και πηγή είναι η δορυφόρη της ροής των δεδομένων. Η μείωση ή η πάυση της ροής δεδομένων θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Και όχι μόνο στον τομέα του διαστήματος. Δεύτερο, αναφερθήκατε στην τεχνολογική πρόοδο. Κανονικά, αν προχωρήσει το Vega C, όπως σχεδιάζεται, θα αντιστοιχεί στο Soyuz το Vega C. Έχουμε ε, εξαντλήσει τη, τη σύμβαση, τα πλαίσια της σύμβασης δεν θα έχουμε πλέον χρήση ρωσικών φορέων, ρωσικών πυράβλων. Και ε, αν το i6 και το ΒΕΓΑ C βγουν στην αγορά εγκαίρως, θα έχουμε ε, πυράβλους εκτόξευσης ε, ευρωπαϊκούς. Και σας ευχαριστώ για την αναγνώρισή σας. Πρέπει να πω ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα του ΤΕΑΣ βάση διανομή στοιχείων του Κοπέρνικος, πληροφοριών του Κοπέρνικος. Η κυρία Βιανκόφσκα, επίτροπός μου, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα την επόμενο, τον επόμενο μήνα και αυτό ήταν απροσδόκητο. Αν δείτε τους βασικούς κανονισμούς που δημιουργούν το Κοπέρνικος, δεν θα δείτε λέξη για την διανομή δεδομένων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις. Δηλαδή, όλα κατασκευάστηκαν για δημόσιους σκοπούς. Και αυτό είναι τρομερό επιτεύγμα. Δεν το πέτυχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απλώς ακολουθήσαμε τελικά τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Συνεργασία ιδιωτικού δημόσιου τομέα τώρα. Χρειαστήκαμε συγκεκριμένη συνεργασία που δεν προβλεπόταν στον οριζοντα 2020 20-2020. Στο νέο κανονισμό θα ενταχθεί ένα άρθρο ούτω ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συνάπτουμε συγκεκριμένες συμφωνίες σύμπραξης στον τομέα του διαστήματος που Εκεί δεν θα, αγοράζονται τα δεν θα αγοράζουμε δεδομένα, αλλά υπηρεσίε. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο μέσω των συμφωνιών αυτών θα δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες, μέσω των συμπράξεων αυτών, αλλά θα δημιουργήσουμε νέες αλυσίδες αξίας. Παράδειγμα, συστήματα υψηλής ανάλυσης λιγότερο από 10% των τροχιών θα χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά επειδή οι δορυφόροι περιστρέφονται πάνω από τους δύο πόλους, 90% της τροχιάς θα εξυπηρετεί και άλλους χρήστες. Πιθανότατα μέσω ιδιωτικής επιχειρήσεως θα πουλούμε τα δεδομένα. Αυτό που θα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα επιτρέπει στις εταιρείε να χρησιμοποιούν αυτούς τους αστερισμούς των δορυφόρων. Δεν θα είναι μόνο συνεργασία ιδιωτικού ε, δημόσιου τομέα για τα στοιχεία του Κοπέρνικος, αλλά θα είναι ένα εργαλείο για την άσκηση βιομηχανικής πολιτικής. Όσον αφορά τα απόβλητα του διαστήματος, συμφωνώ με αυτά που είπατε. Νομίζω ότι το βασικό είναι να αποφύγουμε περαιτέρω αύξηση των αποβλήτων, του αριθμού αυτών. Και στο Γαλιλαίος και στο Κοπέρνικος όλοι οι διαγωνισμοί έγιναν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε όλοι οι δορυφόροι κατασκευάζονται με συστήματα αλλαγής τη τροχιάς. Στο τέλος δηλαδή του προσδοκόμενου κύκλου ζωής του δορυφόρου, τα συστήματα αλλάζουν την τροχιά και ο δορυφόρος καίγεται κατά τη διάρκεια επανεισόδου του στην ατμόσφαιρα. Τέλος, να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι αν υπάρχει ένας τομέας σε παγκόσμιο επίπεδο για την επιτήρηση της γης, παρατήρηση της γης, όπου για μας θεωρήθηκε καταστροφική συνέπεια του Brexit, ε, η καταστροφική συνέπεια στο, στον ε, στο διάστημα. Φανταστείτε ότι πρέπει να παράξω στοιχεία για οποιοδήποτε φορέα της Ευρωπαϊκής Ενώσης όσον αφορά την ασφάλεια στην, στην μάχη να μου λείπουν στοιχεία για ένα κομμάτι της μάχης. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι σχετίζεται με το, νομο... με το διαζύγιο και τις ακολουθούσες διευθετήσεις είναι εκτός αρμοδιότητας. Ο κ. Μπαρνιέ θα ασχοληθεί και η Task Force του άρθρου 50 θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Αλλά για μένα, και αυτή είναι προσωπική άποψη, ε, είναι κοινή λογική ότι όσον αφορά τους δορυφόρους, τα δορυφορικά συστήματα που χρησιμοποιούνται με κάποιο τρόπο, το Ηνωμένο Βασίλειο όπως η Νορβηγία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ε, είναι μέσα από το σύστημα, σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Πέραν του ότι, προφανώς, για κάποια θέματα Πρέπει να βασιζόμαστε σε χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αυτό θεωρείται δεδομένο. Ότι λόγω διμερών διευθετήσεων που υπάρχουν μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας Φερρυπίν στον τομέα της άμυνας μπορούμε να συνεχίσουμε αυτού του είδους τη συνεργασία στο διάστημα. Αυτά. Ευχαριστώ. Thank you, Mr.